Wir Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε παρακαλώ. Έχουμε γεμάτη ημερήσια διάταξη και όπως πάντα έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Σας καλωσορίζω στην ε, συνεδρία της ε, Επιτροπής Πολιτισμού. Ξεκινούμε με το σημείο 1, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Ήδη με email σας έχουμε ανακοινώσει ότι υπάρχει μια αλλαγή στην ε, ημερήσια διάταξή μας. Το αρχικό σημείο 7, την ανταλλαγή δηλαδή απόψεων με την Κομισιόν για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ουγγαρία, θα πρέπει δυστυχώς να την αναβάλουμε. Ε, όχι γιατί βελτιώθηκε καθόλου η κατάσταση στην Ουγγαρία, ε, αλλά επειδή η, την Τετάρτη, την προηγούμενη εβδομάδα, η Κομισιόν δημοσίευσε μια πρόταση για το πρόγραμμα Erasmus Plus, για τα ε, ε, επίγοντα μέτρα για την περίπτωση που έχουμε ε, no deal Brexit στις 29 Μαρτίου. Οπότε πρέπει να συζητήσουμε σήμερα επιγόντω αυτή τη νέα πρόταση τη Κομισιόν και γι' αυτό έχουμε καλέσει εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας παρουσιάσουν αυτή την έκθεση. Αντιρρήσεις υπάρχουν για την αλλαγή αυτή, την τροποποίηση στην ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω κανέναν. Άλλες επιθυμίες για τροποποιήσεις, για συμπλήρωση, για προσθήκη στην ημερήσια διάταξη έχετε. Όχι. Άρα θεωρούμε ότι η ημερήσια διάταξη όπως τροποποιήθηκε εγκρίνεται. Δεν βλέπω να έχει κανείς αντίρρηση. Προχωρούμε. Πάμε στο σημείο 2 της σημερινής διάταξη. Ανακοινώσει τη Προέδρου. Σήμερα έχουμε δύο ερμηνείες της εξή γλώσσες. Γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, πορτογαλικά, τσεχικά, εστονικά, ουγγρικά, πολωνικά, σλοβενικά, βουλγαρικά και ρουμανικά. Όπως πάντα να σα θυμίσω ότι η συνεδρίαση αυτή α, είναι στο διαδίκτυο και επίση να πω ότι τα αποτελέσματα, τη αποφάσεις τη ε, συνεδρίασης των συντονιστών στι 22 Ιανουαρίου 2019, οι οποίες εστάλησαν στις 23 Ιανουαρίου μέσω email στα μέλη της Επιτροπής ε, ε, Πολιτισμού, θεωρούνται πλέον εγκεκριμένε. Εφόσον βεβαίως μέχρι τις 25 Ιανουαρίου δεν είχαν προκύψει αντιρρήσει. Μετά, Πάμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης και είναι οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Και σήμερα ξεκινούμε να ψηφίσουμε την, ε, το σχέδιο ε, έκθεσης. Πρώτο είναι η έκθεση της ε, ε, έκθεσης για τη θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Η συγγήτρια, η συνάδελφος Μιχαέλα Σόντροβα. Έχουμε 332 τροπολογίες. Έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο κατάλογο ψηφοφοριών. Η Μιχαέλα ζήτησε μετά την ψηφοφορία να λάβει το λόγο, οπότε μπορούμε κατευθείαν να περάσουμε στον κατάλογο των ψηφοφοριών. Ε, ελπίζω ότι έχετε όλοι τις κάρτες σας για να ψηφίσετε. Οπότε, ξεκινούμε. Συμβιβαστική πρόταση 1, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 142, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται νομίζω, εξετάζουμε. Λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 142. Πέρας φορέας. 7-7. Απορρίπτεται. Πάμε στην 149. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πάμε πάλι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ρέγγι 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 150. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στην 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στη συμβαστική πρόταση 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ κατά αποχές νομίζω απορρίπτεται αλλά να το δούμε ηλεκτρονικά 158 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας 9-6 απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 163 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έμπλ 26 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω απορρίπτεται, αλλά το ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 8-6. Εγκρίνεται. Πάμε στην 169 και 170. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Έμπλη 27. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχιτη ψηφοφορία. Δεύτερο τμήμα της ΕΜΠΛ 27. Πέρας. 9 ψήφοι υπέρ, 6 κατά. Εγκρίνεται. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 172 σε δύο τμήματα. Η πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται, αλλά ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. η ψηφοφορία. Πέρα. 8 ψήφοι υπέρ, 6 κατά. Εγκρίνεται. 173 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ρέγγι 20. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε στη συμβιβαστική 3, υπέρ. Καλά, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 178, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 179, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 180, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 181, υπέρ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 Απορρίπτεται. 189 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 190 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 204 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Αρχιτή ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τη 204. Πέρας ψηφοφορίας. 7-7. Απορρίπτεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 205. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 206. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται m 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ντεβε 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ψηφίσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίζουμε την ΤΕΒΕ 45. Πέρα ψηφοφορία, 8 ψήφι υπέρ, 7 κατά εγκρίνεται. 207 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έμπλη 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ντεβε 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Είναι πολύ κοντά, κοντινά τα αποτελέσματα. Πέρας ψηφοφορίας. 9 ψήφοι υπέρ, 6 ψήφοι κατά εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην προφορική τροπολογία 3. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Η κυρία Κώστα. Εμείς προτιμούμε την αρχική εκδοχή, πρόεδρε. Ωραία. Αν υπάρχουν πάνω από δύο μέλη της Επιτροπής που είναι αντίθετα, με την προφορική τροπολογία. Θα ψηφίσουμε το αρχικό. Ψηφίζουμε λοιπόν την αρχική τροπολογία. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται στην αρχική τη εκδοχή. ΔΕΒΕ 47. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 209. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 210. Υπέρ. Κατά. απόχέ. Απορρίπτεται. Έμπλ 30. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 211 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 212 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 213 και ρέγγι 22 υπέρ, κατά, αποχές, να το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Geschlossen mit 9 zu 6 abgelehnt. 9 ε, 6 απορρίπτεται. Έμπλη 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 214 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 215 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 216 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 217 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 32, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ντεβε 48, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 218, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ντεβε 49, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έμπλ 32, δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβιβαστική 6, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.24, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέγγι, όχι, πίπτη, 2.25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται, αλλά να το εξετάσουμε. Άρχιτη ψηφοφορία. Geschlossen. Πέρας. Απορρίπτεται. Εμπλ 32 πέμπτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 226. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 227. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 230. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 231 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 236 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 237 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλ 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 243 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 242 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλ 37 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 244 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλ 37 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 245 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλ 37 τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2. Υπάρχουν ενστάσεις, αντιρρήσεις. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν την προφορική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 248. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ψηφίζουμε την 248. Πέρας. Εκρίνεται. 249. Υπέρ. Ηρεμία, ηρεμία σας παρακαλώ. 249 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Μετά έχουμε μία σειρά τροπολογίων τις οποίες δεν θα ψηφίσουμε και θα περάσουμε στην τροπολογία 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Dev 69. Υπέρ. Κατά. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος. Μπάτζ. Μπάτζ 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 256 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 257 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ρέγγι 26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 259 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 260 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μπάντζ 8 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 261 υπέρ. Κατά. Αποχέ. απορρίπτεται. 262 υπέρ. Κατά. Αποχέ. απορρίπτεται. Έμπλη 40 υπέρ. Κατά. Αποχέ. απορρίπτεται. 263 υπέρ. Κατά. Τη 263. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 264. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 265. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Budget 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω πως απορρίπτεται, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται τώρα η ψηφοφορία. Μην κοιμηθείτε παρακαλώ. Όχι ακόμα, δεν ήρθε η ώρα. Πέρας. Απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 266. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 267 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά τη 267. Πέρας. Εγκρίνεται. Χέλγα, πού είναι η κάρτα σου. Την έχεις. Ρέγγι 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 268 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 279 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 285 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 286 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλη 41 τέταρτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 287 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 288. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 289. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 291. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 292. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 290 υπέρ. Κατά. Ξανά υπέρ. Ψηφίζουμε την 290 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 294 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 296 υπέρ. Ναι, 296 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 300 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 301 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 302 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ρέγγι 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 303. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 304. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέγγι 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έμπλη 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 305. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέγγι 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 306. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 1. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 313 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ρέγγι 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 312 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ρέγγι 34 υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέγγι 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 314. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 318. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δέβε 79. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 319 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 320 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 321 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 323 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 322 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 324 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 325 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 326 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έμπλη 44 υπέρ κατά Αποχές θα το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνατε. 10 ψήφι υπέρ, 6 κατά. Έμπλη 45 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έμπλη 45 δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 327 και ρέγκη 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. 327 και ρέγκη 37. Είναι ταυτόσιμες. Αυτές ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται αλλά δεν το είδα πριν. Ρέγγι 38, υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτό θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Μπατζ 10, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έμπλη 45 τρίτο τμήμα και η 328. Όχι. Έμπλη 45 τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 328. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 45 τέταρτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 329 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 330 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Έμπλη 45. Υπέρ. Κατά. Ναι, έμπλη 45. Πέμπτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ούτε το, αυτό ήταν σαφές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την έμπλη 45. Πέμπτο τμήμα. πέρα. Εγκρίνεται. 331 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 332 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έμπλη 45 έκτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Έμπλ 45, 7ο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πάλι την ίδια πλειοψηφία είχαμε, αλλά στο ελέγξουμε. Πέρας. Ναι, 10 ψήφοι υπέρ, 6 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. Έμπλ 45, 8 τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 45, ένα το τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 45, το τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 19, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύε 1, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ντεβε 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ντεβε 3 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έμπλ 2 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία την 43 ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται 8 υπέρ 8 κατά 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ντεβε 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ρέγγι 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω πως εγκρίνεται. Θα το ελέγξουμε όμως. Ψηφίζουμε την 49. Άρχεται η ψηφοφορία. Πολύ γρήγοροι ήμασταν από την αρχή. Παρακαλώ. Δεν ψηφίσαμε όλοι. Τι γίνεται. Την 49 παρακαλώ. Πέρας. 9 ψήφι κατά. Απορρίπτεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ντεβε 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δέβε 6 5. Πρώτο τμήμα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Δεύ 7, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Δεύ 8, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Ντεβ 9, υπέρ. Κατά. Αποχές, νομίζω πως απορρίπτεται. Θα το ελέγξουμε, ψηφίζουμε την DEV 9. Πέρας. Εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Budget 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ντεβε 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έμπλ 8 υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω πως εγκρίνεται. Θα το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την έμπλ 8. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ρέγγι 8 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ντεβε 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έμπλε 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Περνάμε στην έμπλη 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ντεβε 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έμπλη 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύε 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ντεβε 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά εγκρίνεται. Έμπλη 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ντεβε 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ντεβε 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εγκρίνεται, με συγχωρείτε. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 95. Α, με συγχωρείτε. Ναι, ναι, ναι. Λάθος μου στην 96 πάμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ντεβε 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 27. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ρέγγι 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έμπλη 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 116 υπέρ κατά αποχές Δεν ήταν σαφέ. Θα το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 116. Πέρας. Μάλιστα, 13 ψήφοι κατά, 2 υπέρ. Να σηκώνατε τα χεράκια σας παρακαλώ, θα με βοηθήσει. Πού είμαστε τώρα. Ναι, badge 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Dev 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Dev 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Dev 33 υπέρ. Κατά αποχές α, εγκρίνεται. Budget 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 125 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 127 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ντεβε 34 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές θα το ελέγξουμε ψηφίζουμε την 129 πέρας 8 υπέρ 8 κατά απορρίπτεται συμβιβαστική 31 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Ρέγγι 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πως απορρίπτεται αν είδα καλά. Θα το ελέγξουμε όμως. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται καλά που το κοιτάξαμε. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. απορρίπτεται, 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 133 και ρέγγι 18 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. d 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 135 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 138 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Περνάμε στην τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. 14 ψήφοι υπέρ, μία κατά, μία αποχή λοιπόν, με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνεται και συγχαρητήρια στην εισηγήτρια και η Μιχαήλα ζήτησε το λόγο της, ε, τον δίνουμε αμέσω. Ευχαριστώ Πέτρα. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την ε, στήριξη και για την ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ καλή δουλειά που κάναμε, για τη συνεργασία με τους σκιώδε ηγητέ, με την Τερέζα, τη Σίλβια, τη Χέλγκα και επίσης να ευχαριστήσω και το σύμβουλό μας γιατί πραγματικά ήταν ε, δύσκολο το θέμα, αρχικό, αρκετά τεχνικό. Ευχαριστώ τον Λουκά, λοιπόν και την ε, βοηθό μου τη Χριστίνα που είναι εδώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν ε, πολύ καλό το αποτέλεσμα και για τον διαθεσμικό τριμερή διάλογο για τις διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν και προσβλέπω και στην ε, επόμενη καλή μας συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ, ε, Μιχαέλα, για τη δουλειά που έκανες και ευχαριστώ φυσικά και τους σκιώδες συγκητές και τη γραμματεία και όλους όσους συνεργαστήκατε για αυτή την έκθεση. Μπορέσαμε να καταλήξουμε σε καλό αποτέλεσμα. Πάμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία, ε, έγκριση μια γνωμοδότηση, πρόταση του Συμβουλίου, απόφαση Συμβουλίου, με την οποία εξοδοτούνται τα κράτη-μέλη να προσχωρήσουν προ το συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Σύμβαση του Συμβουλίου τη Ευρώπη σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνε και άλλε αθλητικέ διοργανώσει. Η εισηγήτρια, η κυρία Έμα Μακλάρκιν, την οποία δεν βλέπω, προς οπότε προχωρούμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Μία και μόνη τροπολογία, η οποία δεν ήταν αποδεκτή σύμφωνα με τον ιστορικό μας κανονισμό άρθρο 99.1, άρα μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Geschlossen. Πέρας ψηφοφορίας. 16 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά και καμία αποχή. Εγκρίνεται ομόφωνα η έκθεση της κυρίας Μακλάρκιν. Και θα την προωθήσουμε στην καθήλυνα αρμόδια επιτροπή που είναι η ΛΥΜΠΕ. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια, εν τη απουσία της παρόλα αυτά. Κλείσαμε λοιπόν τις ηλεκτρονικές πληροφορίε και πάμε κατευθείαν στο σημείο 5 τη ημερήσια διάταξη πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Η συγκίτρια η κυρία Julie Ward. Οπότε, να πω ότι η προθεσμία για τροπολογίες είναι η 6 Φεβρουαρίου, να το κάνουμε 4. 6 Φεβρουαρίου 4 το απόγευμα. Η προθεσμία αυτή είναι πολύ αυστηρή, το ξέρω, αλλά η ΛΥΜΠΕ έχει τόσο φιλόδοξο πρόγραμμα και έχει προβλέψει την, υψο... την ψηφοφορία στις 21 Μαρτίου. Οπότε... Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να, να καταλήξουμε σε έγκριση σε πρώτη ανάγνωση κατά τη διάρκεια τούτη τη θητεία και η ε, ψηφοφορία θα γίνει στις 11 Μαρτίου σε ειδική σύνοδο στο Συμβούλιο, στο ε, Στρασβούργο, συγγνώμη. Έχουμε ήδη το χρονοδιάγραμμα, έχουμε αφιερώσει το συγκεκριμένο στο συγκεκριμένο θέμα, συγκεκριμένη χρονική περίοδο για να μπορέσει να, συζητηθεί επαρκώς και να γίνει και η ψηφοφορία. Και γι' αυτό θα γίνει σε ειδική σύνοδο στο Στρασβούργο στις 11 Μαρτίου η ψηφοφορία. Πάμε να ακούσουμε τώρα την συνάδελφο Word. Σας δίνω 5-6 λεπτά και να μας παρουσιάσετε την έκθεση. Σας ακούμε. Uh, thank you, Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Καλησπέρα σας. Μετά από κάποιους ε, μήνες συζήτησης ε, στην ΛΥΜΠΕ, η πρόταση κανονισμού για την πρόληψη τρομοκρατικού περιεχομένου ε, online τώρα έχει έρθει προς συζήτηση. Η ΙΜΚΟ εργάζεται επίσης για αυτή την πρόταση ως αρμόδια για γνωμοδότηση επιτροπή. Αυτή η πρόταση θεωρείται προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι θετικό που το Συμβούλιο έχει ήδη συμφωνήσει στη γενική του προσέγγιση υπό την Αυστριακή Προεδρία. Κατανοώ ότι η Κομισιόν σκοπεύει να θέσει εφαρμογή αυτό το κανονισμό όσο γίνεται πιο σύντομα. Στην πράξη, ελπίζουν ότι οι νομοθέτες θα φτάσουν σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση ε, για αυτό το θέμα πριν το πέρα τη θητεία. Αυτό όμω είναι πάρα πολύ φιλόδοξο. Είμαι ευγνώμων στην Επιτροπή που εκπώνησε αυτή την πρόταση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και είμαι ευγνώμων για το ανοιχτό πνεύμα που έδειξαν στην ε, συζήτηση ε, στην DigiCom και τον Επίτροπο και στην King στις προηγούμενες εβδομάδες. Συμφωνούμε επί των αρχών. Ωστόσο, το πρώτο καθήκον που έχουμε ω ευρωβουλευτέ είναι να προστατεύουμε τους πολίτες που υπηρετούμε και εκπροσωπούμε. Και αυτό θα πρέπει να γίνεται μέσω της συνεργασίας και των κοινών αξιών. Τα αίτια της τρομοκρατίας θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στη ρίζα τους και αυτό μπορεί να γίνει αποτελεσματικά μόνο εάν όλοι συνεργαστούν και αν ε, καταβληθεί πανευρωπαϊκή προσπάθεια. Γενικά είναι αποδεκτό ότι ο επιγραμμικός κόσμος παίζει ρόλο κλειδί στο πώς οι τρομοκρατικές ομάδες λειτουργούν, επικοινωνούν, προωθούν και σχεδιάζουν επιθέσεις. Χρειάζεται να αντιμετωπιστεί το παράνομο περιεχόμενο που διαδίδεται online επιγόντως, όμως όχι βιαστικά, ούτε με τίμημα της διάβρωσης της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ασφάλειας. Θα πρέπει να υπάρχουν ε, ε, δυνατότητες ελέγχου και ρήτρε ασφαλείας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως η νομοθεσία θα προστατεύει τις ε, θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα. Νομίζω πως η πρόταση Κομισιόν είναι καλή βάση για συζήτηση, αλλά χρειάζεται αλλαγή στον τόνο. Στην τη σημερινή μορφή το σχέδιο απομακρύνεται από την ισχύουσα νομοθεσία και επιβάλλει νέους κανονισμούς που θα επηρέαζαν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το βασικό κομμάτι του κανονισμού, μάλλον το βασικό θέμα είναι χρονικό, το χρονικό όριο για την ε, διαταγή αφαίρεση. Ξέρω γιατί η Κομισιόν το υποστηρίζει αυτό, γιατί κάποιε στατιστικέ δείχνουν ότι πρώτη ώρα είναι που το παράνομο ε, περιεχόμενο ε, που όταν μάλλον παράνομο περιεχόμενο τοποθετηθεί online ε, προκαλεί τη μεγαλύτερη ζημιά. Όμως είναι σαφές ότι μια διαταγή αφαίρεσης εντός μιας ώρας δεν είναι εφικτή στη, στην πράξη, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν τα κονδύλια ούτε τις δυνατότητες να αντιμετωπίσουν τις διαταγές αφαίρεσης σε τέτοια χρονικά περιθώρια. Πιστεύω πως θα πρέπει να επικρατήσει ευελιξία σε αυτή την πρόταση και να εξασφαλίσουμε ότι το παράνομο περιεχόμενο θα αφαιρείται όσο γίνεται πιο σύντομα και χωρίς ε, καθυστέρηση. Μια σύντομη προθεσμία μαζί με αυστηρά πρόστιμα και χρηματικές ποινές που επιβάλλονται στους παρόχους στο άρθρο 18 σημαίνει πως ε, η πραγματική αφαίρεση δεν θα γίνεται ε, να δεχτεί προσφυγή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περιστάσεις, ο περιπτώσεις μάλλον που θα παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ξέρουμε επίσης ότι κινούμενο περιεχόμενο ή ηχητικό περιεχόμενο μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο από μια ώρα και άρα οι διαταγές αφαίρεσης μπορεί να φτάσουν εκτός ορών γραφείου. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια κοινή οδηγία για όλα αυτά. Όπως όλοι γνωρίζετε, η AMEVS είναι η θεμελιώδη ε, ε, για όλες τις νομοθεσίες σε αυτά τα θέματα και είναι το μεγαλύτερο μας επίτευγμα αυτή τη θητεία. Όμως η Κομισιόν ε, νομίζω πως δεν έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη ε, συνέχεια ανάμεσα σε αυτή την πρόταση και την οδηγία MES e για το οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Δεν αιτιολογείται οποιαδήποτε παρέκκληση ούτε από την οδηγία e-commerce, δηλαδή ηλεκτρονικού εμπορίου και ιδιαίτερα το άρθρο του 15, αλλά ούτε και το 8β που ακριβώς αναφέρεται στην διάδοση παράνομου τρομοκρατικού περιεχομένου online. Δεν είναι συμβατή με την οδηγία ε, ηλεκτρονικού εμπορίου που είναι η νομική αναφορά όσον αφορά την ευθύνη για τους ε, παρόχους ε, φιλοξενίας όπως έχει προβλεφθεί. Μέχρι στιγμής το, το πλαίσιο ευθύνης Απόδοση μάλλον ευθυνών έχει αποδειχθεί επαρκές και έχουν αναπτυχθεί και καλύτερες πρακτικές ώστε να εξασφαλιστεί μια σταθερή και ορθά ρυθμιζόμενη αγορά. Αυτές οι κανονιστικές προσεγγίσεις είναι πολύ σημαντικές για την καταπολέμηση του παρανόμου περιεχομένου ενώ ταυτόχρονα σέβεται τις ε, θεμελιώδεις, ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Στο σχέδιο έχω διαγράψει το άρθρο 6 και πολλοί θα γνωρίζετε ότι στηρίζω τα δραστικά μέτρα στο παρελθόν για νομοθετικού και μη νομοθετικού φακέλους και κυρίως για την παιδική πορνογραφία και εξακολουθώ να στηρίζω τις διασφαλιστικέ δικλείδε. Όμως ε, σε όλα τα μέτρα θα πρέπει να προβλέπεται ο σεβασμός της ισχύουσα ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να δώσει κάποιες νομικές διαβεβαιώσεις διευκρινίζοντα το ε, εκτιμώντας 19 ότι συγκεκριμένα μέτρα δεν θα πρέπει να επιβάλλουν μια γενική ε, ε, υποχρέωση παρακολούθησης, δεν αρκούν ώστε να εγγυηθούν πως δεν θα επιβληθεί καμία γενική υποχρέωση εποπτείας στα κρατημέλη. Επειδή υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι που συνδέονται με την διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου, τα κράτη θα μπορούσαν ενδεχομένως να παρεκκλίνουν από αυτή την αρχή μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, πράγμα που θα οδηγούσε σε μεγάλη αλλαγή στην ισχύουσα νομική προσέγγιση όσον αφορά τους παρόχους φιλοξενίας και του καθεστώτος ε, απόδοσης ευθυνών. Ε, υπάρχει επίσης το θέμα της νομικής εποπτείας όταν πρόκειται για τις διαταγές αφαίρεσης. Υπάρχει ε, ανησυχία ότι είναι οι μόνες αρχές που θα μπορούν να εκδίδουν διαταγές αφαίρεσης αντί για τις αρμόδιες εθνικές δικαστικές αρχές. Θα πρέπει να υπάρχουν ωστόσο δίκαιοι μηχανισμοί ε, διόρθωσης ή αποζημίωσης ή διόρθωσης Διαφορετικά μπορεί να διαλυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και όχι βέβαια οι μεγάλες ε, και βεβαίω η Κομισιόν σκοπεύει αυτό να το ρυθμίσει. Ωστόσο, το άρθρο 18 που ορίζει τι ε, ποινέ για τη συστηματική μη συμμόρφωση θα πρέπει να είναι αντίστοιχα ανάλογε, να μην υπερφορτώσουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, οι οποίε θα πτωχεύσουν μέσω αυτών των ποινών που προτείνει η Κομισιόν. Χρειάζεται βέβαια να επιβληθούν οικονομικές χρηματικές ποινές, όμως η κλίμακα τέτοιων ποινών μπορεί να οδηγήσει ε, ορισμένους ε, παρόχους φιλοξενίας ε, να καταρρεύσουν. Πρέπει να εκτιμηθεί ο αντίκτυπο μια τέτοια νομοθεσία ε, στον κλάδο, ιδιαίτερα στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Η δική μου τροπολογία προτείνει ε, ε, επιβολή ποινών σε εθνικό επίπεδο και βέβαια σε, με, με, σε αναλογία με το μέγεθο των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και την υποδομή cloud και τις υπηρεσίες ε, business to business να εξαιρούνται. Ωστόσο, ήμουν ανέκαθεν υπέρ τη ελευθερία έκφρασης. Ε, εκ των προτέρων ε, προτάσεις ή φίλτρα δεν θα πρέπει να δημιουργήσουν περισσότερη αμφισημία στο κείμενο, γιατί αυτό, κάτι τέτοιο θα έχει επιρροή στην ελευθερία λόγου, αλλά θα είναι και ένας επικίνδυνος δρόμος όσον αφορά την ανάθεση, την εξωτερική ανάθεση της επιβολής του νόμου σε ιδιώτες θα πρέπει να διατηρηθεί ο πλουραλισμός των μέσων ε, και να εξασφαλιστεί η δυνατότητα ε, εκπαιδευτική ε, και η χρήση από τους δημοσιογράφους. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά πόσο ευάλωτοι άνθρωποι μπορεί να πέσουν θύματα των όσων θέλουν να τους βλάψουν και ότι το online περιεχόμενο μπορεί να είναι ιδιαίτερα διαζητικό. Και έχω δει διάφορες πρωτοβουλίες όπου γίνεται προσπάθεια να δοθεί ε, μέσω του ίντερνετ πάλι δυνατότητα στα παιδιά και στους ευάλωτους νέους να εκφραστούν. Ο κανονισμός αυτός από μόνος του δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια. Πρέπει να θαρρύνουμε όλα τα κρατημέλη να επιτείνουν τις επενδύσεις, τις στρατηγικές και τα προγράμματα που στηρίζουν τους νέους, ε, την κοινωνική εργασία, ε, τις πρωτοβουλίες από ριζοσπαστικοποίηση, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να ευθυγραμμιστεί με επίσημη ενημέρωση και την ανεπίσημη παιδεία όσον αφορά την γνώση χρήσης των μέσων μαζικής ενημέρωσης καθώς ε, και συνεργασία με τα δίκτυα από ριζοσπαστικοποίηση. Συγγνώμη, δεν έχω πολύ ακόμα, λέει ο Μιλήτρια, ενώ η Πρόεδρος τη διακόπτει και συνεχίζει να διαβάζει ακόμη πιο γρήγορα. Ενώσει των νέων και εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να μπορέσουν να αντισταθούν στα ακραία μέτρα μέσω περισσότερης εκπαίδευσης. Τέτοιες πρωτοβουλίες συχνά συμβαίνουν σε, μικρές, σε μικρή κλίμακα Άρα λοιπόν στηρίζω γενικά τα διάφορα στοιχεία και επιχειρήματα αυτής της πρότασης. Κυρία Γουόρντ, σας παρακαλώ, λέει η Πρόεδρος. Συνεχίζει η κυρία Γουόρντ, Θα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν οι απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας πριν αυτό να γίνει κοινοτική νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδότησης. Πάμε τώρα στους σκιώδεις συζητητές αν βλέπω καλά, μόνο δύο είναι παρόντες. Οπότε ξεκινούμε με τη Χέλγα Τρούπελ. Ευχαριστώ, Τζούλη, ευχαριστώ, Πέτρα. Again, a big question of conflict of goals. We want... Και πάλι το θέμα είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία στο διαδίκτυο, κυρίως όταν είναι ξεκάθαρο ότι είναι τρομοκρατικό το περιεχόμενο και συνδέεται με, την, ε, με τα όσα έχουμε ορίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως τρομοκρατία. Από την, την ίδια στιγμή όμως δεν έχουμε και ξεκάθαρο ορισμό της τρομοκρατίας, οπότε είναι αρκετά περίεργος ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να προσπαθήσουμε να ρυθμίσουμε το περιεχόμενο. Και από την άλλη έχουμε και το θέμα της έκφρασης τη ελευθερία της έκφρασης. Να ξεκινήσω με ένα ερώτημα για τα φίλτρα ε, uploading. Ε, σε αντίθεση με σένα, Τζούλη, εγώ νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια, ένα ξεκαθάρισμα τη οδηγία ε, του ηλεκτρονικού εμπορίου, γιατί αν έχουμε το safe harbor εντάξει, τον ασφαλή λιμένα, αν κάνουμε ό,τι κάναμε και για την οδηγία για τις ε, οπτικοακουστικές υπηρεσίες, νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα. Το θέμα δεν είναι να έχουμε μόνο ελευθερία στο ίντερνετ, αλλά να δούμε και τι κάνουν όντω οι πάροχοι υπηρεσιών. Το άρθρο 13 της οδηγίας για το copyright είναι ε, ούτως ή άλλως ε, θέμα και ηθικής αλλά και ε, δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Οπότε, όπως ξέρετε, εγώ είμαι υπέρ του άρθρου 13 της οδηγίας copyright γιατί δεν είναι υποχρεωτική η, το φιλτράρισμα για το upload, αλλά για την Κομισιόν νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ πιο, πιο επικίνδυνο, γιατί εδώ προσπαθούμε να περιορίσουμε το περιεχόμενο. Οπότε καταλαβαίνω αυτό που λες, Τζούλη, πρέπει όντω να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε σχέση με το τι θα κάνουμε και πρέπει να δούμε ποιο είναι ο ορισμός της τρομοκρατίας. Έχουμε αξιολόγηση αντικτύπου, τις οδηγίες για την τρομοκρατία. Αν έχουμε, εγώ θα την ήθελα να τη δω πριν προχωρήσουμε και επίσης χρειάζεται ένας ξεκάθαρος ορισμός των αρχών που είναι, αρχέ, που είναι υπεύθυνες και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να μπει και, στην, και στις τροπολογίες, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε κράτος δικαίου, γιατί αλλιώς ε, ιδιωτικοποιείται η ευθύνη. Εκχωρούμε την ευθύνη σε ιδιωτικές εταιρείε να λάβουν δράση. Και αυτό από μόνο του, από πολιτική πλευρά, δεν νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει λύση. Και σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε χρόνο. Κατανοώ ότι υπάρχει άμεση ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία στο διαδίκτυο, αλλά τώρα να, να κάνουμε γρήγορα με ένα τόσο σημαντικό ε, θέμα για τη ρύθμιση του περιεχομένου μέσα σε λίγες εβδομάδες, δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη συζήτηση και με το νέο κοινοβούλιο για συνολικά το θέμα της ρύθμισης περιεχομένου. Χρειαζόμαστε ξεκάθαρους ορισμούς, χρειαζόμαστε να ορίσουμε τι είναι, ο, ποιος είναι ο ρόλος των δικαστών, πώς μπορούμε να πληρώσουμε για να έχουμε σωστή δικαιοσύνη, πώς μπορούμε να βρούμε τα κονδύλια για τη δικαιοσύνη. Και πρέπει να δούμε τι γίνεται και online, τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Είναι επίγον το θέμα, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, ακόμη και αν είμαστε ήδη έτοιμοι τώρα, να λύσουμε το πρόβλημα της, ε, του, της κατανομής των ρόλων. Η Κομισιόν προσπαθεί να βρει ένα σωστό ορισμό, προς το παρόν δεν νομίζω ότι έχει καταφέρει, δεν έχει ολοκληρώσει τη δουλειά αυτή και δεν νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε για να λύσουμε αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα με τον λάθος τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το να καταπολεμηθεί το τρομοκρατικό περιεχόμενο online είναι απαραίτητο. Το είδαμε πρόσφατα στη Λιβύη, όπου αντέλασαν οι τρομοκράτες ε, απόψεις στο Facebook ε, με πλήρη τιμωρησία. Ωστόσο, θα πρέπει να ορίσουμε καλύτερα το τρομοκρατικό ε, περιεχόμενο ενώ πρόκειται ας πούμε για άρθρο εφημερίδας εκεί φαίνεται να είναι λίγο υπερβολικό θα πρέπει να το τρομοκρατικό περιεχόμενο δεν έχει να κάνει με ελευθερία λόγου, δεν έχουμε κάνει τέτοια συζήτηση σε πολύ πιο επίμαχα ζητήματα. Και αυτό ενώ η ύπατη αρμοστία των, Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει εκφράσει σοβαρέ επιφυλάξει για το γερμανική σχετική νομοθεσία, για παράδειγμα. Επίση, λυπούμε που δεν μπορούμε να κάνουμε μια πραγματική συζήτηση για την πολιτική λογοκρισία που γίνεται όλο ένα και πιο ύπουλα στα κοινωνικά δίκτυα όπως το Twitter, ε, κάποιες φορές μέσω αλγορίθμων που επιτρέπουν να κρύβονται ορισμένα πολιτικά περιεχόμενα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Μαρίτερες Τερές Χιμένες έχει το λόγο. Εκ μέρους λοιπόν της οργανωσής μας θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεση, η οποία έχει αρκετά ισορροπημένη προσέγγιση στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα γίνονται σεβαστά σε ό,τι φορά την ε, αφαίρεση ε, περιεχομένη απομάκρυνση προσώπων. Ωστόσο, χρειάζεται να ε, τονίσουμε το θέμα της, του χρονοδιαγράμματος και της πίεσης του χρόνου. Γι' αυτό, λοιπόν, πρέπει να το τονίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάποιες παρατηρήσεις και από μένα θα ήθελα να κάνω τώρα, να σας πω πως ε, πολεμήσαμε με την Επιτροπή ε, ΛΥΜΠΕ για να καταφέρουμε να καταρτήσουμε γνωμοδότηση επίσης ε, σύμφωνα με το άρθρο 54 και να συμμετέχουμε και εμείς λοιπόν ε, εδώ και το χρονοδιάγραμμα της ΛΥΜΠΕ το έκανε σχεδόν αδύνατον για μας να καταφέρουμε να εργαστούμε και νομίζω πως δεν μπορούμε να δεχτούμε ε, τον τρόπο που έχουν προτείνει να δουλέψουμε. Να σας ε, πω ειλικρινά πως είμαι εκνευρισμένη, διότι εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν είχε ζητήσει νομοθετική λύση του θέματος, θα προτιμούσα να το εξετάσουμε σε μια άλλη χρονική περίοδο και όχι στο τέλος της κοινοβουλευτικής ε, θητείας όπου εμείς ε, βρισκόμαστε πλέον ε, σε, σε, στην τελική ευθεία δεχόμαστε μεγάλες πιέσεις και δεν μπορούμε λοιπόν να εργαστούμε με τρόπο ικανοποιητικό σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν μπορούμε να εξετάσουμε το θέμα, να το συζητήσουμε, να δούμε με προσοχή το θέμα του διαχωρισμού μεταξύ των θεμελιωδών δικαιωμάτων από τη μία και του νομικού περιεχομένου από την άλλη. Επίσης, ε, με την Σαμπίνα Φερχάιεν ήμασταν συνεισηγήτριες ε, και έχω να πω πως ε, είναι πολύ δύσκολο. Δεν μας βοήθησαν καθόλου, ιδιαίτερα σε το φορά τους πρώτερους ελέγχους ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται όντως για τρομοκρατικό περιεχόμενο εδώ λοιπόν εμποδίζεται η άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Περιορίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι πάροχοι υπηρεσιών ε, έχουν υποβαθμιστεί σε παιδονόμους, σε ρήφιδες. Και εκείνοι πρέπει να αποφασίσουν λοιπόν και να κρίνουν αν ένα περιεχόμενο είναι απειλητικό ή πιθανώς ε, τρομοκρατικό στην ε, οδηγία για, τα, για τις ε, υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ε, πάλι τα ίδια έγιναν, πάλι τα ίδια συζητήσαμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει μια πρόταση η οποία κατά τη γνώμη μου δεν είναι δυνατόν να εξεταστεί και να διηγηθούμε σε μια σύμφωνη γνώμη. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε πάλι σε αυτή την άποψη της Κομισιόν λοιπόν, ε, και βασίζομαι πάνω σε διάφορες διατάξει τη οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Γι' αυτό λυπάμαι πάρα πολύ για το ότι μας έχει ασκηθεί τόσο έντονη πίεση χρόνου, ε, ακριβώς όπως την εποχή που συζητούσαμε για το περιεχόμενο που σχετίζεται με παιδική πορνογραφία και είπαμε ότι ναι φυσικά πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά, ναι φυσικά πρέπει να ε, προστατεύσουμε από πιθανές τρομοκρατικές, ε, τρομοκρατικό περιεχόμενο όπως στην προκειμένη περίπτωση, όμως πρέπει να γίνει ε, ένας διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτό που αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και σε αυτούς που χρήζουν προστασία από την άλλη. Αυτή λοιπόν η συζήτηση θα έπρεπε να γίνει, αλλά δυστυχώς στην προκειμένη περίπτωση δεν προλαβαίνουμε, δεν έχουμε το χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Τζούλη, η οποία μας παρουσίασε μια τόσο ισορροπημένη έκθεση, η οποία ε, φυσικά βάζει στο προσκήνιο τα θεμελιώδη δικαιώματα και από ε, την άλλη τονίζει ότι αυτά είναι ε, δικαιώματα τα οποία πρέπει αδιαφημισβήτητα να προστατεύονται. Είναι μια θέση η οποία νομίζω πως ε, δεν θα είναι δύσκολο να ε, γίνει αποδεκτή και από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Αυτά ήταν τα προσωπικά σχόλια. Και να σας πω επίσης ότι δύο συνάδελφοι έχουν ζητήσει το, λόγιο, το λόγο, ο κύριος Ντρογεύσκη και ο κύριος Μόρκανο και η Σίλβια Κώστα λοιπόν. Μετά θα λάβει το λόγο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Στρογεύσκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω από κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Λοιπόν, ε, σε ό,τι αφορά την στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής Λίμπερ, να πω τα εξή ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συστήσει μια ειδική υποεπιτροπή ε, με το όνομα ΤΕΡ για την, ε, για την εξέταση θεμάτων σχετικών με την τρομοκρατία. Υπήρξαν όμως πάρα πολλά προβλήματα με την όλη διαδικασία, με την εξέταση της έκθεσης εννοώ. Χρειάστηκε πάρα πολύ χρόνος και η έκθεση αυτή εγκρίθηκε μόλις ε, πρόσφατα. Η Επιτροπή Λίμπε λοιπόν δεν είχε αρκετό χρόνο και ως εκ του αποτελέσματος δεν είχαμε ούτε εμεί αρκετό χρόνο να εξετάσουμε την έκθεση. Γιατί εδώ δεν γίνεται λόγος για την ελευθερία στο διαδίκτυο, αλλά για θέματα τρομοκρατίας. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο έχει να κάνει με απειλές, σωματικές απειλές, σωματικό κίνδυνο των ε, πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε εδώ να ισορροπήσουμε τα πράγματα ανάμεσα στις ευαισθησίες από τη μία της ε, Julie Ward, της εισηγήτριας, και από την άλλη της, ε, των, των πιθανών τρομοκρατών. Πρέπει λοιπόν να διατηρηθούν αυτές οι πολύ λεπτές ισορροπίες. Επίσης, ε, προβλέπεται μια εξαίρεση για συγκεκριμένες ομάδες δημοσιογράφων για τους οποίους δεν θα ισχύουν περιορισμοί στην αναζήτηση. Επίσης, και οι κατηγορούμενοι έχουν δικαιώματα. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Η ειδική λοιπόν επιτροπή για την τρομοκρατία προσπάθησε να προσαρμόσει τους ορισμούς καταλήλως, όμως ε, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το έργο της. Θα πρότεινα λοιπόν να υπάρχει μεν ε, κάποια λογική συνέχεια, μια συμφωνία με αυτές τις ευαισθησίες, όμως να μην υπερβούμε τις αρμοδιότητές μας, ε, διότι διαφορετικά ε, θα εργαστούμε υπέρ των τρομοκρατών. Μην ξεχνάτε επίση ότι οι τρομοκράτε εργάζονται πάρα πολύ γρήγορα και α, όταν κάποιο ε, θέλει μία ώρα για να απομακρύνει τρομοκρατικό περιεχόμενο, αυτή η ώρα είναι πάρα πολύ χρόνο. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει δυνατότητα γρήγορης διαδικασίας. Θα προτιμούσα λοιπόν λύσεις οι οποίες είναι εντός των αρμοδιοτήτων μας και να διατηρηθεί η ισορροπία δυνάμεων εδώ. Σας ευχαριστώ. Κύριος Μόργανο. Σας ευχαριστώ. Εγώ ήθελα να θυμίσω τα εξή. Καταρχά, ευχαριστώ την Τζούλη για τη δουλειά που έκανε, για την απόπειρα να συνδυάσει τι διάφορε ευαισθησίε και σωστά τα υπογράμμισε αυτό. Ωστόσο, θα πρέπει να πω ειλικρινά πω έχω την εντύπωση πω κάποιε ανησυχίε που αναφέρθηκαν είναι κάπω υπερβολικέ. Τι σημαίνει αυτό. Άλλο είναι να βρούμε την σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την ελευθερία ε, και τη σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και άλλο είναι να εξετάσουμε το αντικείμενο που έχουμε ενώπιόν μας. Είναι ένας κανονισμός, δηλαδή άμεσα εφαρμοστέως, ο οποίος πρέπει να αφορά την, ε, τον εντοπισμό και την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου online. Και εδώ η μεταβλητή του χρόνου έχει σημασία. Δεν είναι αδιάφορο η χρόνη αντίδραση, Γιατί το υπογραμμίζω αυτό, γιατί το βασικό θέμα είναι, ε, νομίζω πως η ε, κάθε φορά που γίνονται επιθέσεις, ε, η τελετουργία κάθε φορά ε, πια δεν έχουν ε, χρόνο. Ε, τι βρισκόμαστε να κάνουμε, τι. Εκφράζουμε τη λύπη μα, αλλά το θέμα είναι μαζί με την Κομισιόν και το Συμβούλιο πρέπει να δώσουμε απάντηση. Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν ε, ε, κάνουμε το καθήκον μα, που δεν είναι μόνο ηθικό καθήκον, είναι και θεσμικό καθήκον απέναντι στου συμπολίτε μα. Αν λοιπόν εγώ μέσω του ίντερνετ βάζω και λέω πώς μπορεί κανείς να κατασκευάσει μια βόμβα, δεν θα πρέπει να προσεχθεί επειδή είναι ελεύθερη ενημέρωση ή είναι κάτι άλλο. Όταν βλέπω ας πούμε ότι νέοι Σουηδοί ε, αποκεφαλίστηκαν και το βάζω εγώ στο ίντερνετ, μα αυτό τι είναι, ελευθερία έκφρασης. Δηλαδή θεωρώ πως είναι ένα πολύ σημαντικό ανθρώπινο πρόβλημα. Πού θέλω να καταλήξω. Εάν ε, η κατάσταση ήταν δυνατόν να λυθεί, δεν θα είχαμε ενώπιόν μας σε αυτή την κατάσταση. Τα όσα έγιναν τώρα, μέχρι τώρα, δείχνουν ότι δεν έχουμε κάνει αρκετά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα παρεύουμε ή όχι. Μέσος δρόμο, μέσο η οχι μεσος δρομο μεσο η δεν υπάρχει. Και ε, ε, αν εδώ αφαιρέσω την σαφήνεια των κανόνων και των ποινών, των αποτρεπτικών ποινών, τότε θα είναι ένας κανονισμός που δυστυχώς δεν έχει νόημα. Άρα λοιπόν, άλλο είναι να λέμε πως δεν είναι όλες οι πραγματικότητες όντω να φτάσουν στην πράξη. Οκ, ναι, το καταλαβαίνω. Όταν η Τζούλη αναφέρεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα λοιπά και ότι δεν θα τα καταφέρνουν, αλλά ορισμένα θέματα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πως οι πλατφόρμες μπορούν να τα κάνουν, γιατί διαφορετικά τα... Ε, ήταν ένα άλλο είδος παρέμβασης. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει σε συνεννόηση με, τους αρμόδιους, με τα αρμόδια όργανα θα πρέπει να κάνουμε τα κατάλληλα βήματα για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Αν μετά από 20 χρόνια φανταζόμαστε πως βάση των όσων κάνουμε είναι η οδηγία e-commerce, εγώ συμφωνώ με την Τρούπελ γι' αυτό. Το είπα και το έχω δηλώσει και σε άλλες περιστάσεις όταν έγινε λόγος για VMS και τα λοιπά. Προσοχή, ο η τρομοκρατία είναι πολύ σοβαρό θέμα. Η ασφάλεια είναι πολύ σοβαρό θέμα και τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι και η προστασία της ασφάλειας όλων. Εντάξει, μακρηγόρησα πάντω είναι θέματα που δεν μπορούμε να τα λύσουμε ε, λέγοντας άστο για την άλλη φορά. Άμα ο καθένας λέει άστο για την επόμενη φορά, ε, τότε θα πρέπει να αναλάβουμε και ο καθένας τις πολιτικές μας ευθύνε. Ευχαριστώ. Πρέπει να σας ζητήσω κάτι, παρόλο που είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η συζήτηση, να μην κάνουμε αυτά που ε, θα μας ε, κατηγορούσαν ότι προσπαθούμε να ε, καλύψουμε ή να προστατεύσουμε τους ε, τρομοκράτες. Πρέπει να βρούμε τη σωστή ευαίσθητη αυτή η ισορροπία. Το λέω, το ξαναλέω, ας είμαστε πολύ προσεκτικοί. Η κυρία Κώστα έχει το λόγο. Ε, Μάλιστα, είναι δύσκολη η ισορροπία που πρέπει να προστατευσουμε τους τρομοκρατες πρεπει να βρουμε τη σωστη ευαισθητη αυτη ισορροπια το λεω το ξαναλεω ας ειμαστε Ευχαριστώ την Τζούλη γιατί μίλησε για το ποια είναι ε, ε, η ισορροπία από την πλευρά της Επιτροπής ε, Πολιτισμού. Συμμερίζομαι ίσως κάποια από αυτά που είπε, ότι δηλαδή είναι τόσο σύντομο το χρονικό διάστημα, όπως έλεγαν και οι άλλοι συνάδελφοι. Έχουμε εδώ και έχουμε μια εις βάθος συζήτηση, δεν έχουμε κάνει μάλλον εις βάθος συζήτηση, γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα. Μα ζητήσανε με ψήφισμα να παρέμβουμε ήδη, ζητήσαμε μάλλον με ψήφισμα από πέρσι την παρέμβαση. Δεν έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να εμβαθύνουμε. Ίσως θα ήταν καλό κάπως περισσότερο να σε περιοριστούμε, όπως ε, να περιοριστούμε στις αρμοδιότητές μας και να μην μπούμε στα άρθρα τα οποία αφορούν ε, θέματα ορισμών που ε, είναι θέματα της ΛΥΜΠΕ. Δεύτερον, θεωρώ σε αυτή την πρόταση ότι γίνεται μια απόπειρα να οριστεί το τρομοκρατικό περιεχόμενο. Μπορεί να πούμε ότι ναι, δεν είναι ίσως κατάλληλο, αλλά για πρώτη φορά ορίζονται όλα αυτά. Ίσως αυτό το οποίο είναι πιο περίπλοκο να είναι ότι ίσως θα πρέπει να περιοριστούν κάπως οι ορισμοί, γιατί είναι πολύ ευρύς αυτό μπορούμε να το δούμε. Όμως ορισμοί υπάρχουν για το ποιο, τι είναι το περιεχόμενο. Δεν είναι αλήθεια ότι έχει μείνει ε, αόριστο. Έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις στη συνάδελφο Word. δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για παρόχους υπηρεσιών ε, εντός της Ένωσης, γιατί ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάροχοι υπηρεσιών που είναι, έχουν έδρα σε τρίτες χώρες, αλλά λειτουργούν ε, μέσα στην Ένωση. Κάτι ακόμα δεν μπορούμε να πούμε μόνο για την ε, δικαστική αρχή που αυτή μπορεί όντως να παρέμβει όποτε θέλει, αλλά στις διάφορες αρχές, αρχές τηλεπικοινωνιών κτλ. Και έπειτα το να λέμε ότι πρέπει να περιοριζόμαστε σε εκείνους τους ε, προμηθευτές παρόχους υπηρεσιών που απευθύνονται σε ένα γενικό ακροατήριο. Προσοχή! Όχι μόνο είναι ο πάροχος υπηρεσιών που απευθύνεται στο γενικό κοινό, στο ευρύ κοινό, αλλά έχουμε και το darknet. Έχουμε εκείνο το, το darknet που είναι πολύ επικίνδυνο. Το 6 και το 9 τώρα, τα άρθρα 6 και 9 είναι, είναι δύσκολα. Δεν μπορούμε να, να διαγράψουμε το 6 και τη σύνδεσή του με το 9, που είναι αυτό που αφορά τις εγγυήσει και τη δυνατότητα προσφυγής. Νομίζω πως κάτι τέτοιο θα ήταν ότι θα σήμερα να ξεπεράσουμε την ισορροπία. Συμμερίζομαι και αυτό που είπε ο Λουίτζι Μόργανο και η κυρία Τρούπελ για το e-commerce. Ήταν δική μας καθυστέρηση αυτή εδώ τη θητεία. Η επόμενη θητεία θα πρέπει να το αντιμετωπίσει, γιατί και το άρθρο 14 και 15 του e-commerce εγγυώνται ότι πρέπει να υπάρχει ευθύνη, αλλά όχι σε δύο περιπτώσεις όταν πρόκειται για παρανομία και όταν δεν ενεργήσουν άμεσα για να αφαιρέσουν. Εδώ πρόκειται για τρομοκρατικό περιεχόμενο και πρέπει κάπως να ε, ξεπεράσουμε την ερμηνεία που δίνει η οδηγία e-commerce. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να απαντήσω λίγο στην ε, συζήτηση που προέκυψε από αυτή την πρόταση. Πρέπει όντως να εξορροπήσουμε το ε, δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης με την ασφάλεια. Ε, εδώ προσπαθούμε να συζητήσουμε πάνω στην ισορροπία μιας πρότασης με την οποία πολλές φορές έχουμε προβλήματα. Βεβαίως θέλουμε να υπάρχει ελευθερία έκφρασης, αλλά φυσικά πρέπει να διασφαλίσουμε και την ασφάλεια, κυρίως στον τομέα του διαδικτύου. Πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει κανείς τους σωστούς συμβιβασμούς. Η Πέτρα μίλησε για τις ε, οπτικοακουστικές υπηρεσίες και εδώ μιλούμε για περιεχόμενο και νομίζω ότι έχουμε βρει καλή λύση. Αλλά βεβαίως υπάρχει όντως ε, ε, αντίσταση. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι η λύση που έχουμε βρει είναι σωστή. Γιατί βασικά διασφαλίζεται το δικαίωμα της ζωής. Αυτό λέει και η Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και νομίζω ότι όλα, αυτό, το, αυτή, αυτό το δικαίωμα του να ε, δημοσιεύονται όλα στο ίντερνετ πρέπει να το δούμε και υπό το πρίσμα της ασφάλειας. Εκεί που απειλείται η ζωή πρέπει αυτό το, το δικαίωμα να περιορίζεται. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και υπό το πρίσμα των θεμελιδών δικαιωμάτων αλλά και υπό το πρίσμα της ασφάλειας των πολιτών. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, να προσθέσουμε και εμείς κάποια σχόλια. Καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε για την πολύ καλή και πολύ σοβαρή συζήτηση που κάνετε για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ε, ζητούμε συγγνώμη που ε, φτάνει στο τέλος της θητείας του Κοινοβουλίου σας η πρόταση αυτή, αλλά όπως είπατε όλοι είναι σοβαρό το θέμα αυτό και επειδή ακριβώς είναι σοβαρό χρειαζόμαστε και κάποια α, ε, τεκμηρίωση κάποια τεκμηρίωση που θα, δημιουργούν, που θα δημιουργεί ένα σύνδεσμο μεταξύ περιεχομένου στο ίντερνετ και της ριζοσπαστικοποίησης μεμονωμένων πολιτών και βεβαίως τρομοκρατικών επιθέσεων. Και υπάρχει ριζοσπαστικοποίηση online σε κάθε περίπτωση τρομοκρατικής ενέργειας από το 2015 και μετά. Χρειάζεται λοιπόν πραγματικά στέρεη τεκμηρίωση, απόδειξη. Γι' αυτό χρειάστηκε να γίνει αυτή η πρόταση για να ξεπεράσουμε τα όσα έχουμε πετύχει τα τελευταία δύο χρόνια σε θελούσια βάση. Υπάρχει μια στιγμή όπου κάνει κανείς μια σωστή αξιολόγηση για το κατά πόσο μπορεί όντως να λειτουργήσει σε θελούσια βάση ή αν χρειάζεται να επιβάλλει κάτι. Αυτή την απόφαση έπρεπε να λάβουμε εμείς και πραγματικά μας ενθάρρυναν και όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ως προς αυτό. Σας ευχαριστώ επίσης που το λαμβάνετε τόσο στα σοβαρά. Ευχαριστούμε για την αρχική έκθεση και όχι μόνο για αυτή, αλλά και για τα σχόλια όλα που μόλις ακούσαμε. Θεωρούμε ότι όντως υπάρχει σοβαρή ευκαιρία τώρα να συμφωνήσουμε επί εύλογου συστήματος που θα έχει αποτελέσματα αλλά που δεν θα διακυβεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και την ελευθερία της έκφρασης. Η συγκήτρια πολύ σωστά είπε στο σχέδιο εκθεσής της ότι υπάρχουν πολλά θεμελιώδη σημεία, είναι ο ορισμός ένα εξ αυτών και θεωρούμε ότι η πρόταση που ήδη υπάρχει στο σχέδιο έκθεσης πηγαίνει προς την σωστή κατεύθυνση να ξεκαθαρίσει, να περιορίσει ακόμη περισσότερο αυτό που ακριβώς θέλουμε να στοχεύσουμε. Τώρα, για, το, για την εντολή απόσυρσης του περιεχομένου και, την, το που προερχεται στο σχεδιο κειμενου εγγραφου οραματιστεί. Όπως είπατε και εσείς, θεωρούμε ότι το θέμα της, ε, των εντολών απόσυρσης ε, πρέπει να ξεκαθαριστεί ε, σαφέστατα. Δεν μπορούμε αυτό να το αφήσουμε στα χέρια του οποιοδήποτε. Αυτό θα πρέπει να οριστεί, να καθοριστεί ξεκάθαρα, να ελέγχεται, να, να ξέρουμε ποιες θα είναι οι αρχές που θα το κάνουν. Αλλά το να το αφήσουμε και πάλι μόνο στα, στα χέρια ενός δικαστή πάει πολύ μακριά. Πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα που θα επιτρέπει αρχές που θα εποπτεύονται να κάνουν αυτή τη δουλειά, να εκδίδουν δηλαδή εντολέ απόσυρση. γιατί ακριβώς είναι πολύ ισχυδείς οι περιπτώσει που προκύπτουν στα διάφορα κράτη-μέλη. Θεωρούμε ότι αυτά τα προληπτικά μέτρα είναι απολύτως απαραίτητα και έγινε η συζήτηση για το θέμα της ε, συνάφειας με την οδηγία ε, του ηλεκτρονικού εμπορίου και στο ιστορικό της Κομισιόν, αλλά και με τα κράτη-μέλη όταν το ε, Συμβούλιο καταλήξε στη γενική του προσέγγιση. Οπότε θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε κάποια προληπτικά μέτρα και υποχρεώσεις πολύ φιλόδοξα για τον κλάδο, χωρίς όμως να εμποδίζουμε ή να διακυβεύουμε τις βασικές αρχές που υπάρχουν στην ε, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο ή σε άλλα νομοθετικά κείμενα, μερικά εκ των οποίων τα γνωρίζετε πολύ καλά. Τώρα, για τις ασφαλιστικές δικλείδες, στο σχέδιο κειμένου, στο σχέδιο έκθεσης, βλέπουμε ότι όντως είναι ένα πολύ σημαντικό. Ένα τελευταίο, τελευταίο θα πω, Πρόεδρε. Υπάρχει, γίνεται μια προσπάθεια να υπάρξει ακόμη καλύτερος ορισμός αυτών των ασφαλιστικών δικλείδων. Το καλωσορίζουμε, το χαιρετίζουμε και θα είμαστε στο πλευρό σα σε κάθε περίπτωση για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε την περαιτέρω και να παράσχουμε την τεχνηρίωση που χρειάζεστε για τι διάφορε πτυχέ που άπτονται αυτού του σχεδίου ε, νομοθεσία. Σα ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Νόμιζα ότι ε, θα ήταν το να το αποφασίζουν όλο αυτό οι δικαστικοί, ότι είναι βασικό πυλώνα τη δικαστική ανεξαρτησία, αλλά προσπαθώ ίσω να έκανε και λάθο. Τζούλη, έχει το λόγο. Ε, ελάχιστο χρόνο θα σου δώσω. Έχουμε ήδη ξεπεράσει το πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πάω έτσι κι αλλιώ στην Επιτροπή Λίμπε για να ψηφίσω για μια άλλη έκθεση ω αναπληρωματικό μέλο. Ε, νομίζω πω η συζήτηση είναι πολύτιμη εδώ. Χρειάζεται σαφήνεια και αυτό είναι τόσο σημαντικό ε, σε ένα θέμα στο οποίο παρατηρώ πως υπάρχει έλλειψη σαφήνειας για ό,τι έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα. Θα πρέπει να ε, μιλήσουμε για παράνομο τρομοκρατικό περιεχόμενο, αλλά τι σημαίνει παράνομο. Ε, τι σημαίνει πιθανά επιβλαβές. Τι σημαίνει αυτό. Με την ε, Γιούλια Ρέντα συζητούσαμε με τον εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν την περασμένη εβδομάδα και μας είπε ότι είναι πολύ εύκολο ας να βρει κανείς στο διαδίκτυο πώς μπορεί να φτιάξει ένα ε, πολύ τοξικό δηλητήριο. Ρικίνη. Είναι μια γνώση που βρίσκεται ελεύθερα στο διαδίκτυο και ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ε, το τι συμβαίνει, την ε, διάδοση και την ε, ύπαρξη της πληροφορία, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι να εκπαιδευτούμε για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πιθανές απειλές. Και σε αυτό ακριβώς το θέμα υπάρχει τέτοια έλλειψη σαφήνειας που δυσχεραίνει το έργο μας και τη θέση μα απέναντι στις άλλε επιτροπές. Και αυτό είναι πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω και εσένα Πέτρα και τους συναδέλφους που πολέμησαν σκληρά έτσι ώστε να αποκτήσουμε και εμείς αρμοδιότητα για αυτό το θέμα. Και εμείς στην Επιτροπή Πολιτισμού υπερασπιζόμαστε τι πολιτικέ ελευθερίε. Βασικά όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να το κάνουμε. Εμείς όμως ε, υπερασπιζόμαστε τις ε, πολιτικές ελευθερίες ε, πάνω και πέρα από όσα κάνει η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μεν η κατανόηση στις αξίες, στις θεμελιώδει αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως εγώ θέλω να γίνει συζήτηση ουσιαστική και να συζητήσουμε σημαντικά θέματα. Σίγουρα θα έπρεπε να έχει συζητηθεί το θέμα βέβαια πολλά χρόνια πριν, 4-5 χρόνια πριν, έτσι δεν είναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρεπτόντος να σας ενημερώσω ότι δεν ε, δρούμε σε, ένα, σε περιβάλλον ανομίας, υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν πλαίσια και έχουμε ένα κείμενο να ψηφίσουμε το οποίο ακριβώς ε, για αυτό το θέμα μιλά. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι 6 Φεβρουαρίου στις 4 το απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, ε, για το οποίο δυστυχώς έχουμε μόνο μισή ώρα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Όμως θα περάσουμε τώρα στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης, μια μελέτη που ζήτησε η Επιτροπή μας, την οποία ανέθεσε στο θεματικό τμήμα το... για την επιστήμη και τον επιστημονικό γραμματισμό ως εκπαιδευτική πρόκληση. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω τον Ντάλιμπορ Στέρν Άντελ, από το Ινστιτούτο Δημόσιας Πολιτικής και Διαχείρισης της Λιθουανίας, ο οποίος με κατόπιν ε, ανάθεσης της ε, Επιτροπής μας θα μας παρουσιάσει την ε, μελέτη, η οποία δεν είναι ακόμα έτοιμη, όμως ήδη παρουσιάζει τα πιο ουσιαστικά σημεία. Η μελέτη θα ολοκληρωθεί και θα δημοσιευθεί το τέλος ε, Φεβρουαρίου. Θα ήθελα να καλωσορίσω λοιπόν τον κύριο Στέρν Άντελ, να τον ευχαριστήσω που ήρθε και να του δώσω το λόγο για την παρουσίαση της μελέτης, η οποία για μας είναι πάρα πολύ σημαντική, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της ε, πολιτικής συζήτησης για την εκπαίδευση, με το οποίο μας, ε, η οποία η πολιτική μας απασχολεί σε αυτήν την θητεία έντονα. Σας παρακαλώ λοιπόν να μην ξεπεράσετε τα 10 λεπτά, έτσι ώστε να έχουμε χρόνο και για συζήτηση. Έχετε λοιπόν το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Ντάλιμπορ Στέιναντελ από το Ινστιτούτο Μελετών στην, ε, στο Βίλνιο, της ε, Λιθουανίας. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν ε, τα αποτελέσματα της μελέτης μας. Είμαι ένας από τους συντάκτες της μελέτης αυτής λοιπόν και η περίληψη της με παρουσίασης είναι διαθέσιμη σε εσάς. Στι ερχόμενε εβδομάδες λοιπόν θα δημοσιευθεί και η μελέτη στο σύνολό τη. Είναι λοιπόν μια ανασκόπηση της ε, βιβλιογραφίας για την, ε, τον επιστημονικό γραμματισμό και την ε, χρήση στην πράξη σε πολιτικές και σε πλαίσιο εκπαιδευτικό. Το θέμα αυτό εξετάζεται στο πλαίσιο της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων, των fake news, της διάδοσης ε, ψευδών ειδήσεων εσκεμένα. Ιδιαίτερα σε θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος όπως η υγεία, η περιβαλλοντική πολιτική, κάτι το οποίο τους ε, περασμένους μήνες έχει γύρει πολλά ερωτηματικά. Εξετάζεται λοιπόν και η παραπληροφόρηση και οι επιπτώσεις που έχει στην ικανότητα των πολιτών ε, να ε, αξιολογούν την πληροφορία και καταστάσεις ε, αυτές. Επίσης, στην μελέτη γίνεται μια ανασκόπηση των διαθέσιμων δεδομένων σχετικά με τον επιστημονικό γραμματισμό στον ευρύτερο πληθυσμό και ασχολούμαστε με τις ε, εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που μπορούν να βελτιώσουν την ενημέρωση του πληθυσμού ο επιστημονικός γραμματισμός στη βιβλιογραφία έχει διάφορες, ε, διάφορους ορισμούς. Είναι η ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς επιστημονικά ζητήματα ως σκεπτόμενος πολίτης. Ε, σύμφωνα με αυτό είναι, αυτός ο ορισμός του ωσα ε, στο πλαίσιο των τεστ PISA. Ο επιστημονικός γραμματισμός όμως μπορεί να εξεταστεί και από ένα ευρύτερο πλαίσιο ως κοινωνική ως κοινωνικό φαινόμενο και εδώ εξετάζονται η κριτική σκέψη, η ενασχόληση με τα κοινά και άλλες πτυχές της ε, δημόσιας ζωής που μπορούν να έχουν σχέση με τον επιστημονικό γραμματισμό. Επίσης, λοιπόν, βλέπουμε ότι τούτος είναι ένα, μια έννοια η οποία η οποία σχετίζεται και με πολλούς άλλους τομείς που επηρεάζουν την κριτική σκέψη του ατόμου. Τώρα, από τους ορισμούς που έχουμε εξετάσει και από την βιβλιογραφία, μπορούμε να κάνουμε τις εξή συστάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεδομένη στις περιορισμένες αρμοδιότητας το, της ε, Κομισιόν και της αποκλειστικής αρμοδιότητας των κρατών μελών για θέματα εκπαίδευσης να ε, συνδράμει στην ε, σωστή εφαρμογή του πλαισίου για τον γραμματισμό και για τη βελτίωση της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής των κρατών μελών. Όπως είπα και πριν, σε αυτήν την εποχή παραπληροφόρησης είναι πολύ σημαντική ε, η αναγνώριση της ε, αλήθειας. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε πώς διαδίδονται οι ψευδείς πληροφορίες και πώς αυτό είχε άμεσες επιπτώσεις σε διάφορα θέματα όπως αμβολιασμός, για παράδειγμα, ή παραπληροφόρηση σχετικά με την ασφάλεια κάποιων εμβολίων και πώς αυτό οδήγησε στην εξάπλωση ορισμένων νόσων όπως ε, όπως η Λαρά. Επίσης, ε, εξετάζονται και οι προκαταλήψεις ε, του κοινού από την άποψη της ψυχολογίας όπου παρατηρείται πως ε, ο άνθρωπος αναζητά πληροφορίες οι οποίες επιβεβαιώνουν τις δικές του πεπιθήσεις. Επίσης εξετάζεται και το φαινόμενο όπου όταν ένας άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με πληροφορίες οι οποίες ε, διαφωνούν με τις προσωπικές του πεπιθήσεις, αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις και στην ουσία ενισχύει την, ε, άποψη, την αντίθετη άποψη του ατόμου. Επίσης εξετάζονται οι διάφορες πλατφόρμες ε, που δημιουργούν αυτό που λέμε αντίλαλο, δηλαδή όπου παρουσιάζεται μια πληροφορία η οποία επίσης επιβεβαιώνει μια ε, πρώτερη υπεποίθηση, λανθασμένη ενδεχομένως. Και αυτό, όπω σα είπα και πιο πριν, είχε άμεσε επιπτώσει σε διάφορε συζητήσει με θέμα τον εμβολιασμό, την κλιματική αλλαγή, οδήγησε σε ε, συνένεση βασισμένη σε παραπληροφόρηση. Παρά το γεγονός ότι στο θέμα της κλιματικής αλλαγής ο άνθρωπος είχε άμεση επιρροή στην κλιματική αλλαγή και Εξετάζεται επίση το πλαίσιο στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει, να βοηθήσει ας πούμε σε θέματα σχολικής εκπαίδευσης, σε θέματα ευαισθητοποίησης, όπου η διασταύρωση στοιχείων είναι πολύ σημαντική και πρέπει να ε, διδάσκεται. Εξετάζεται λοιπόν η ψευδής πληροφορία ο, κατά κάποιο τρόπο σαν ένα ιός κατά του οποίου οι πολίτες πρέπει να εμβολιαστούν. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες προσεγγίσεις που βασίζονται σε μία προσέγγιση σε τρία στάδια. Δίνεται έμφαση στο γεγονός, στα στοιχεία και όχι στις ε, ψευδείς πληροφορίες. Για παράδειγμα, ας πούμε, κλιματική αλλαγή, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι έχουν ε, επηρεάσει το περιβάλλον. Ε, αυτό ε, εξετάζεται σε αντιδιαστολή με το μύθο, ας πούμε, ότι ναι, η έκρηξη ενό φεστίου μπορεί επίσης να αυξήσει τα επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα. Διαψεύδονται λοιπόν αυτές οι λανθασμένες πληροφορίες, ότι ναι, μεν το ηφαίστειο επηρεάζει, αλλά όχι τόσο όσο η ανθρώπινη δραστηριότητα. Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις στην ε, βελτίωση του επιστημονικού γραμματισμού. Αυτός δεν προσμετράται στα τεστ πιζα Επίσης παρατηρούμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι μαθητές δεν ακολουθούν σπουδές που έχουν να κάνουν με την επιστήμη. Μόνο το 15% των φοιτητών ακολουθούν τέτοιους κλάδους σπουδών. Υπάρχουν βέβαια διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη, τις εξετάζει και αυτή η έκθεση. Σε ορισμένες χώρες υπάρχει λοιπόν ε, χαμηλή, χαμηλό ενδιαφέρον ανάμεσα στα, στους 15χρονους μαθητές για επιστημονικά θέματα ε, αναλύονται οι έρευνες του Ευρωβαρόμετρου όπου φαίνεται πως τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεν μια θετική στάση των πολιτών απέναντι σε διάφορα θέματα περιβαλλοντικά, για παράδειγμα. Βλέπουμε ότι το 90% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρεί πως η κλιματική αλλαγή είναι σοβαρό ζήτημα. Και οι συστάσεις μας, βάσει της έρευνας και των στοιχείων που έχουμε εξετάσει, είναι η λήψη πρωτοβουλειών που θα βελτιώσουν τον, τον επιστημονικό γραμματισμό. Αντλούμε από τις έρευνες του Ευρωβαρόμετρου και η σύσταση είναι να υπάρχει καλύτερη εκπαίδευση έτσι ώστε να αναγνωρίζονται και να εντοπίζονται ε, οι αιτίες της παραπληροφόρησης. Μετά, Εξετάζουμε την εκπαιδευτική πολιτική στα κρατημέλη και τι γίνεται για να ενισχυθεί ε, ο επιστημονικός γραμματισμός. Βλέπουμε πως δεν υπάρχει μια κοινή προσέγγιση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα πλαίσιο και διάφορα μέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει τα κρατη σε αυτό το σκοπό. Εξετάζεται η διδακτέα ύλη και έμφαση που δίνει κάθε κράτος μέλος στην επιστήμη, αλλά και στην εφαρμογή της στην πράξη. Επίσης, εξετάζονται τα αποτελέσματα, όπου παρατηρούνται μεγάλες διαφορές από κράτος σε κράτος. Και βλέπουμε πως υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις ε, προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών. Από τη μία έχουμε δηλαδή τον ε, εκπαιδευτικό στις φυσικές επιστήμες, ο οποίος ε, οδηγεί τους μαθητές στο αποτέλεσμα μέσω πειραμάτων και από την άλλη βλέπουμε την ε, παραδοσιακή διδασκαλία. Βλέπουμε όμως ότι η διδασκαλία βασισμένη στο πείραμα οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα, γιατί ο μαθητής αποκτά μία πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση του ζητήματος που εξετάζει κάθε φορά. Μετά, θα μπορούσαμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσουμε το Erasmus Plus και άλλα παρόμοια προγράμματα τα οποία θα ενισχύσουν ε, την, ε, τις, ε, τα προσόντα και τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών ακριβώς γιατί η επιτυχία της, ε, στον, στον επιστημονικό γραμματισμό στηρίζεται στους εκπαιδευτικούς. Αυτά λοιπόν ε, εν ολίγη ήταν μια πολύ πολύ γρήγορη και σύντομη περίληψη και θα χαρώ πολύ να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Όντως, ε, χρησιμοποίησατε πολύ έξυπνα το χρόνο σας. Και βεβαίω φαντάζομαι ότι περιμένουμε όλοι και την τελική εκδοχή της έκθεσης. Κοιτάζω γύρω-γύρω στην αίθουσα να δω αν υπάρχουν παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Η Χέλγα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Χαίρομαι που μπορούμε να κάνουμε έτσι μια μικρή παρέμβαση πριν έρθουν τα τελευταία στοιχεία για να έχουμε και μια ιδέα του τι κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και το θέμα είναι λίγο θέμα ενημέρωσης, διαφωτισμού. Είναι σημαντικό, οι επιστήμες πάντα συνδέονται με το διαφωτισμό στην ευρωπαϊκή ιστορία και πραγματικά τίνουμε, κυρίως αν δούμε και τις δημόσιες συζήτηση που γίνεται για τους εμβολιασμούς ας πούμε, έχουμε το στρατόπεδο που είναι υπέρ των εμβολιασμών και των, ε, της ε, ιατρικής που βασίζεται στα αποδεικτικά στοιχεία, στο οποίο ανήκω και εγώ, και το άλλο στρατόπεδο που αμφισβητεί όλα τα στοιχεία. Ο επιστημονικός λοιπόν χρωματισμός νομίζω ότι έχει πάρα πολύ να κάνει με το πώς αντιλαμβανόμαστε τους επιστήμες, την επιστή, τους επιστήμονες, την επιστήμη και την ελίτ, γιατί και η ελίτ είναι κάπως συνδεδεμένη με την επιστήμη. Πρέπει κανείς να έχει σπουδάσει πολύ, να έχει πολύ σοβαρό υπόβαθρο για να καταλάβει περί τίνος πρόκειται όταν μιλούμε για επιστήμες. Και το βλέπουμε ότι στις σύγχρονες κοινωνίες έχουμε πολλούς ανθρώπους που μιλούν κατά τον ελίτ εξ ονόματος των πολιτών. Και εσείς από ό,τι καταλαβαίνω προτιμάτε την προσέγγιση που λέει ότι οι μαθητές, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν με τα επιστημονικά πεδία γιατί έτσι μόνο θα καταλάβουν και θα εμπλακούν στην όλη διαδικασία, θα συμμετάσχουν στη διαδικασία των επιστημονικών ευρημάτων και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη η μελέτη σας. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η Μαρή Τερέζ. Ευχαριστώ πολύ αυτή την έκθεση. Ε, θα περιμένουμε τα, τελευταία, τα τελικά σας πορίσματα και πώς βλέπετε εσείς τη σχέση που έχουν ορισμένα πράγματα ή μάλλον ε, επιθύσεις ε, που δημιουργούνται για την, με την επιστήμη σε σχέση με τον λαϊκισμό. Ε, ορισμένες φορές ο λαϊκισμός ε, ή διάφορες απόψεις που επικρατούν όπως ας πούμε υπάρχουν εκστρατείες ε, εναντίον των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ή εναντίον συνόλων πολιτών που, που υποτίθεται βασίζονται στην επιστήμη. Μια, ένα επιχείρημα ας πούμε, που ε, ε, ε, ίσχυσε για τη γλυφοσάτη ήταν ότι ένα εκατομμύριο άνθρωποι είχαν υπογράψει εναντίον της γλυφοσάτης. Μα αυτό δεν είναι επιχείρημα που ένας πολιτικός μπορεί να το χειριστεί σε σχέση με το αν ναι ή όχι μπορεί να εγκριθεί ένα χημικό, μια χημική ουσία ή όχι. Και άλλη μια ερώτηση που θέλω να υποβάλω είναι ότι ε, κάποιες ε, μαρτυρίες δείχνουν ότι οι προσωπικές ιδεολογικές διαφορές οδηγούν και σε ε, διαφορές επιστημονικού τύπου. Δηλαδή, οι φιλελεύθεροι και οι συντηρητικοί συνηθίζουν να αμφισβητούν επιστημονικές απόψεις. Για να αποφύγουμε αυτό το την κομματική, της κομματικό διχασμό, θα έπρεπε ίσως να κάνουμε εκπαιδευτικές δραστηριότητες με εκπροσώπους όλου του πολιτικού φάσματος. Εσείς έχετε κάποια ιδέα για το πώς θα μπορούσαμε να το πετύχουμε αυτό. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπίλτ. Pardon. Μάλιστα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ κύριε. Είναι κρίμα που δεν είχαμε γνωρίσει τα πορίσματα αυτή τη έρευνα λίγο νωρίτερα για ένα τόσο κρίσιμο θέμα όσο είναι η επιστημονική κουλτούρα και επειδή αναφέρατε πολύ ενδιαφέροντα θέματα όπω ε, τα εμβόλια, οι κλιματικέ αλλαγέ. Είναι κρίσιμο επίση γιατί προχωράμε προ το 2020 και είναι εντυπωσιακό ότι οι στόχοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά τη σχολική αποτυχία δεν θα επιτευχθούν η αποτυχία στις επιστήμες ήταν 22,20 το 2015 και ε, μεγάλη ήταν η αύξηση σε σχέση με το 2012. Αναφέρεται διάφορους παράγοντες, αλλά ένα ε, φαινόμενο που είναι ταμπού στη Γαλλία είναι η διείσδυση του θρησκείας στα σχολεία. Το θέμα έχει μελετηθεί στη ΣΥΠΑ όπου κάποιες αντιδραστικές ομάδες έχουν μεγάλη δραστηριότητα. Φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στις ε, ε, ε θρησκευτικές πεπιθήσεις και τις επιστήμες. Στη Γαλλία ο καθηγητής Ζαν Πατίστη Παναφιέ έχει μελετήσει τους μουσουλμάνους φοιτητέ, ε, σπουδαστέ, οι οποίοι αρνούνται να ε, παρακολουθήσουν τα μαθήματα, ας πούμε, για την εξέλιξη του ανθρώπου. Έχετε μελετήσει αυτό το θέμα και πώς ε, εσεί πιστεύετε ότι μπορεί να ξεπεραστεί το θέμα της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην επιστήμη και τον φονταμενταλισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μας δίνετε την ε, ευκαιρία να έχουμε μια εικόνα της δουλειάς σας. Δύο ερωτήματα έχω. Υπάρχουν διάφορες οπτικές ε, ε, για το πώς μπορεί κανείς να προσλάβει, να κατανοήσει τα επιστημονικά ευρήματα, πώς μπορεί να κάνει από μόνος του επιστημονική δουλειά, αλλά υπάρχει και το ερώτημα πώς μπορούμε να φέρουμε κοντά την επιστήμη στους πολίτες, ακόμα και σε αυτούς που δεν ε, μπορεί να, που μπορεί να μην έχουν ε, ψηλή εκπαίδευση ε, για να την καταλάβουν. Τι γίνεται ως προς αυτό, να καταλάβουν δηλαδή ακόμα και βασικές αρχές της επιστήμης. Εδώ, Εδώ νομίζω ότι το θέμα του επιστημονικού γραμματισμού πρέπει να το α, δουλέψουμε στα διάφορα επίπεδα. Η επιστημονική κατανόηση πρέπει να έρθει κοντά στους πολίτες, όχι κατά ανάγκη αυτούς που την έχουν σπουδάσει μόνο. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να γίνει αυτό ε, και με θέσεις και με αντιθέσεις βεβαίως ε, που εκπροσωπούνται σήμερα από το και με να το πούμε με απλά λόγια. Το να μιλούμε έτσι όλοι πολύ επιστημονικά ίσως να, είναι, να καθιστά πιο δύσκολη την κατανόηση. Οπότε ίσως αυτή την προσέγγιση θα πρέπει να την, έχουμε, να την βάλουμε στον, ε, στην όλη συζήτηση, να προωθήσουμε την επιστήμη, αλλά όχι μόνο την επιστήμη προ χάρη τη επιστήμη και των επιστημόνων ή των ανθρώπων που έχουν σπουδάσει, αλλά ανθρώπου που μπορεί να μην έχουν τελικά τόσο υψηλή εκπαίδευση. Ευχαριστώ. Η κυρία Κώστα τελευταία. Σα ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες, ε, την ενδιαφέρουσα έρευνα και για την πρόκληση που ακούστηκε όσον αφορά τα ερωτήματα και τις πιθανές ε, συστάσεις. Η επιστημονική κουλτούρα είναι κυρίως αυτή που δίνει μια μεθοδολογία, δηλαδή μια επιστημονική προσέγγιση στην οποία καταρτίζεται ο άνθρωπος. Αυτό ισχύει τόσο για τις ανθρωπιστικές όσο και για τις θετικές επιστήμες. Είναι σύνολο ε, αυτό. Η επιστημονική σκέψη είναι μεθοδολογία προσέγγισης και όχι μόνο ε, πλαίσιο των θετικών επιστήμων. Θέλω να καταλάβω να συμφωνείτε. Ε, έπειτα, πιστεύω πως υπάρχουν αντιφάσεις, το είπατε και εσείς μάλιστα, στο πλαίσιο της έρευνάς σας. Έχω την εντύπωση λοιπόν πως υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε μια στάση που πιο ενδιαφέρουσα να πάρει κανείς περισσότερη επιστημονική ε, κουλτούρα, ενώ αντίθετα μειώνονται οι δεξιότητες. Οι, οι επιστημονικές ε, δεξιότητες λόγω των μεγάλων διαφορών στα σχολικά συστήματα στην Ευρώπη. Έχετε κάποιες εξηγήσει γι' αυτό, δηλαδή καλές και κακές πρακτικέ. Και το τελευταίο θέμα είναι πώ θεωρείτε στις περίφημες 8 δεξιότητε κλειδιά που πρέπει να έχει κάθε πολίτη. αν εσεί πιστεύετε ότι έχουμε ε, ότι θα πρέπει να σκεφτούμε κάτι διαφορετικό όσον αφορά την απόκτηση επιστημονικών γνώσεων. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας ζητήσω να προσπαθήσετε να απαντήσετε εντός 5 λεπτών. Θα προσπαθήσω λοιπόν να απαντήσω σε όσο το εντών περισσότερες ερωτήσεις. Μέτρησα τις ερωτήσεις. Αρκετές είναι. Να ξεκινήσω από το θέμα του εμβολιασμού. Όπως και για το πόσο ευθύνεται το άνθρωπος για την κλιματική αλλαγή, ούτε εδώ έχει γίνει συζήτηση, έχει υπάρξει διάλογος για την ε, ασφάλεια ορισμένων εμβολίων. Για παράδειγμα, το εμβόλιο MMR, το τριπλό, για την Ιλαρά... και δεν θυμάμαι δυστυχώς για ποιες άλλες ασθένειες. Υπήρχε ένα πέπλο μυστηρίου, υπήρχε παραπληροφόρηση. Είχε δημοσιευτεί μάλιστα και ένα άρθρο βασισμένο σε λάθος πληροφορίες, το οποίο κατηγορούσε το εμβόλιο ε, ότι ήταν ε, αναποτελεσματικό χωρίς να βασίζεται σε στοιχεία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να βελτιωθεί η αντίληψη ε, των ε, πολιτών. Και εδώ γυρίζουμε πάλι στην εκπαίδευση. Χρειάζεται λοιπόν να ενημερώσουμε, να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές για το τι σημαίνει επιστημονική συνένεση, για το πώς αποδομείται ένας ε, μύθος, μία ψευδής πληροφορία. Τώρα, για την ελιτιστική προσέγγιση που αναφέρατε, βλέπουμε κάποια θετικά παραδείγματα. Για παράδειγμα, το πώς η επιστήμη μπορεί να γίνει δημοφιλής, πώς η επιστήμη γίνεται αγαπητή. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την εκπαίδευση, όχι μόνο των ε, παιδιών αλλά και των ενηλίκων, διότι βλέπουμε πολλές φορές πως η παραπληροφόρηση για επιστημονικά ζητήματα γίνεται εκτός ε, σχολικού περιβάλλοντος, γίνεται μεταξύ ενηλίκων. Γι' αυτό είναι σημαντικό λοιπόν να γίνουν προσπάθειες εκλαΐκευσης της επιστήμης από διάφορα μουσεία, διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ε, τα οποία θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο εγχείρημα αυτό. Επίσης, η ανοιχτή επιστήμη, όπου δηλαδή οι επιστήμονες θα βγουν έξω από τα εργαστήρια, ανάμεσα στους πολίτες, θα προωθήσουν τις μελέτες τους και ίσως αυτό βοηθήσει να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στην επιστήμη και τον ευρύ πληθυσμό. Επίσης, η διαφάνεια των αποτελεσμάτων είναι εξίσου σημαντική για να επανέλθω ε, στο ερώτημά σας για την ε, κλιματική αλληλή. Χρειάζεται λοιπόν να δοθεί μια διαφάνεια ιδιαίτερα στις μεθόδους επαλήθευσης ε, που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες. Εδώ λοιπόν όσοι χαράσουν πολιτική έχουν πολύ και σημαντική δουλειά μπροστά τους. Μετά, αντίκτυπος ε, στην ε, αντίληψη, στις ε, απόψεις των πολιτών. Πράγματι, ορισμένοι ενισχύουν τις πεπιθήσεις τους με την δημοσίευση στοιχείων αντίθετων προς αυτές. Και εδώ πάλι θα επιστρέψω στην επιστημονική συνένεση, όπου πρέπει να προωθήσουμε αυτό το γεγονό ότι όλοι οι επιστήμονες συμφωνούν τα τελευταία 200 χρόνια η δράση του ανθρώπου επηρέασε το ε, ε, κλίμα. Χρειάζεται λοιπόν και πάλι να γίνουν προσπάθειες ε, να αποδομηθούν αυτές οι αναλήθειε, αυτός ο μύθος για το ότι ο άνθρωπος δεν ευθύνεται για την κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις βέβαια, αλλά είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι τα στοιχεία δείχνουν πως υπάρχει μία κατεύθυνση. Δεν πρέπει να δίνουμε βάση στις ψευδείς ειδήσει, διότι αυτές ε, υπονομεύουν την επιστημονική αλήθεια, τα επιστημονικά στοιχεία. Αυτό είναι κάτι στο οποίο συμφωνούν περισσότεροι επιστήμονες. Νομίζω πως κάλυψα τα περισσότερα σημεία των ερωτησεών σας. Προσπάθησα να το κάνω εγκάρση, αλλά δεν, βλέπ, δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση, όμω θα απαντήσω με τα χαρά και σε άλλες. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα για να μας παρουσιάσετε τη μελέτη που σας αναθέσαμε. Αν υπομονούμε να διαβάσουμε την τελική μορφή της μελέτης, σας ευχόμαστε καλή συνέχεια λοιπόν και σας τονίζω άλλη μια φορά ότι περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον διότι η μελέτη σας θα βοηθήσει και στη δική μας δουλειά. Θα μας βοηθήσετε με τα ευρήματά σας λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. So, das geht hier heute Schlag auf Schlag. Frau Eriksen, mögen Sie zu mir kommen? Λοιπόν, κυρία Έριξον, ελάτε στο Προεδρείο, γιατί θα περάσουμε στο νέο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης, στην ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση των μέσων ε, έκτακτης ανάγκης ε, και το πώς το Brexit θα επηρεάσει ορισμένα προγράμματα όπως το Erasmus+. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκεται ενώπιον μας η κυρία Έριξον. Έχει ξανάρθει στην Επιτροπή θα μας παρουσιάσει λοιπόν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, από την περασμένη εβδομάδα. Θεωρώ πως ε, θα πρέπει να φροντίσουμε ότι σε περίπτωση ενός σκληρού Brexit όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό ή έχουν άδεια να μεταβούν στο εξωτερικό από τις 29 Μαρτίου και μετά ή να σπουδάσουν, να κάνουν πρακτική οτιδήποτε άλλο στο Ηνωμένο Βασίλειο να έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές στην πρακτική τους ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να προσέξουμε για να μην φύγει κατά τα πόδια μας, λοιπόν, και για αυτό το σκοπό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μία πρόταση την περασμένη εβδομάδα και η κυρία Έριξον θα μας την παρουσιάσει αμέσως τώρα. Αυτό είναι και ένα θέμα το οποίο θα εξετάσουμε και στη συνάντηση των ε, συντονιστών, διότι πρέπει να εργαστούμε ταχύτατα έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ε, μία άποψη, σε μία πρόταση, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε πώς θα προστατευτούν οι πολίτες και από τις δύο πλευρές σε περίπτωση ενός σκληρού Brexit. Κύριε Έριξον, έχετε το λόγο και σας ευχαριστούμε άλλη μια φορά για την πρότασή σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την εισαγωγή σας. Να σας πω κάποια βασικά στοιχεία της ε, πολύ πρόσφατα υιοθετηθής σας, ε, ε, μάλλον του πολύ πρόσφατα υιοθετηθέτους κανονισμού για την συνέχιση των δραστηριοτήτων εκμάθησης, εκπαίδευσης στα περίπτωση του hard Brexit και γενικώ στην περίπτωση της, του, της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κανονισμός αυτός προσπαθεί να δημιουργήσει κάποια μέτρα προληπτικά για να αποφύγουμε μεγάλη αναταραχή. Για προγράμματα όπως το Erasmus Plus, προγράμματα μετακίνησης, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει στην, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία για να γίνει αυτό. Ε, είναι κομμάτι των, των προσπαθειών που κάνει η Κομισιόν να έχει γενικότερα μέτρα αναδίπλωσης, οπότε θεωρούμε ότι είναι μια άμεση λύση σε ένα άμεσο πρόβλημα αυτή που προτείνουμε. Και για να έχουμε έτσι κάποια αριθμητικά στοιχεία. Προς το παρόν, το, προς τη στιγμή της αποχώρησης, μπορεί να έχουμε περίπου 14.000 συμμετέχοντες της Ευρώπης των 27 στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα έχουμε περίπου 7.000 ε, Βρετανούς σε, στην Ευρώπη των 27. Ε, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία, αυτό σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες του Erasmus Plus θα πρέπει να διακόψουν τελείως τι δραστηριότητε αυτέ τη ε, εκμάθηση ε, μέσα από το πρόγραμμα κινητικότητα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι πραγματικά καταστροφικό για του φοιτητέ αυτού, αλλά και για τι ε, χώρε που του φιλοξενούν, για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, προφανώ για του φοιτητέ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διακόψουν τι σπουδέ του και να επιστρέψουν στη χώρα του. Μπορεί να χάσουν τα ακαδημαϊκά του credits, μπορεί να χάσουν το εξάμεινό του. Οπότε θα είναι πραγματικά καταστροφικό. Ο, το σχέδιο αυτό κανονισμού έχει μόνο τέσσερα άρθρα, είναι πολύ σύντομος ο κανονισμός αυτός και θέλει να προστατεύσει τους συμμετέχοντες από αυτή την καταστροφή. Είναι σημαντικό να προστατεύσουμε λοιπόν τις τρέχουσες διαδικασίες κινητικότητας τη στιγμή της αποχώρησης και είναι σημαντικό επίσης να καλύψουμε και αυτούς που βρίσκονται στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω Εράσμους και προγράμματος χρηματοδοτηθέντος από το από το Εράσμο και αυτούς που είναι Βρετανοί και σπουδάζουν σε άλλη χώρα. Οπότε έχουμε ας πούμε έναν Γάλλο σπουδαστή ε, στο Λονδίνο μέσω Εράσμους και έχουμε και έναν Βρετανό ο οποίος κάνει την ε, πρακτική του ε, σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Επίσης είναι σημαντικό να πούμε ότι οι συμμετέχοντες θα ε, ολοκληρώσουν την περίοδο αυτή της κινητικότητας και θα, συνεχίσουν να ε, λαμβάνουν τη χρηματοδότηση που πρέπει. Οπότε, σε σχέση με το τι καλύπτει ο κανονισμός. Το πεδίο εφαρμογής του δείχνει ότι εφαρμόζεται για όλους τους, ε, για όλες τις του Erasmus στα πλαίσια του, της δράσης 1 του κανονισμού Erasmus Plus που ξεκίνησανε πριν από την ημερομηνία αποχώρησης. Οπότε έχουμε την ε, δραστηριότητα κινητικότητα έτσι όπω ορίζεται αυτή στον ε, κανονισμό. Έχουμε ε, φοιτητέ, άτομα που κάνουν πρακτική, μαθητεία, φοιτητέ, μαθητέ σε επαγγελματικά προγράμματα, κινητικότητα νέων σε άτυπη και μη επίσημη εκπαιδευτική δραστηριότητα, εθελοντέ, κινητικότητα εργατικού δυναμικού για κατάρτιση και κινητικότητα ατόμων που δουλεύουν σε οργανισμούς νεολαίας. Ε, αυτό είναι το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Επίση σημαντικό είναι ότι εφαρμόζεται σε συμμετέχοντες από και προς όλα τα χώρε προγράμματο όλες τις, χώρες προγράμματος ε, του Erasmus Plus και το Ηνωμένο Βασίλειο και βεβαίως το έχουμε και την... Ε, το Λίχτενστάιν, την Νορβηγία, την Ισλανδία, την Φίρομ και την Τουρκία. Επίση σημαντικό είναι ε, ότι δεν είναι ε, ε, προϋπόθεση η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στον προϋπολογισμό του 2019 και επίσης δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, εκπνοής. Η δραστηριότητα δηλαδή, η κινητικότητα μπορεί να συνεχιστεί μέχρι να ολοκληρωθεί. Βεβαίως η μεγαλύτερη διάρκεια είναι 12 μήνες, όπως ξέρουμε. Επίσης, ξέρουμε ότι πρέπει να το γνωστοποιήσουμε αυτό σε όσους είναι σε αυτό το πρόγραμμα κινητικότητας, οπότε θα ενημερώσουμε όλους τους συμμετέχοντες για όλα αυτά μέσω των εθνικών σημείων επαφής, που είναι ε, οι υπηρεσίε Erasmus Plus σε κάθε χώρα και όπως ξέρετε, ε, ξέρετε καλά τον κανονισμό άλλωστε, πρέπει να περάσουμε από τη διαδικασία συνομοθεσίας, οπότε είναι προ συμφέρον όλων να αποφύγουμε αυτέ τι καταστροφικέ συνέπειε. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε την κατανόησή σα για το πολύ συγκεκριμένο αυτό πρόβλημα και ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε ε, γρήγορα και απρόσκοπτα να εγκριθεί ο κανονισμό αυτό για να αποφύγουμε ακριβώ αυτέ τι καταστροφικέ συνέπειε για όλους αυτούς τους ε, συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus+. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ένα ερώτημα μου ήρθε τώρα στο νου τι γίνεται με τους συμμετέχοντες στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντισμού στα πλαίσια ας πούμε, αυτό, αυτών που δουλεύουν στο ε, σώμα αλληλεγγύης. Ε, και αυτοί μάλλον πλήττονται. Δεν ξέρω, αυτή η επικάλυψη μεταξύ σώματος αλληλεγγύης και σώματος εθελοντών ε, καλύπτεται από τον κανονισμό σας. Μήπως έχετε ξεχάσει κάποια ομάδα, μήπως τους ξεχάσατε αυτούς. Και κοιτάζω και γύρω-γύρω να ξεκινήσω με τη Σαμπίνε ως συντονίστρια. Ένα νομικό ερώτημα έχω. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συντάσσουμε ένα νομικό κείμενο για το τι θα γίνει με τους συμμετέχοντες σε, αυτούς τους, σε αυτά τα προγράμματα. Αν υπάρξει hard Brexit, η Βρετανική πλευρά δεν θα δεσμεύεται πια από την ε, νομοθεσία που θα ψηφίσουμε εμείς. Οπότε πώς θα, πώς εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι 7.000 ε, Βρετανοί ε, που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι 14.000 Ευρωπαίοι που είναι στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορέσουν να συμμορφωθούν με την νομοθεσία που θα υπάρχει γιατί είναι δίκοπο μαχαίρι. Υπάρχει κάποιο είδους ανταλλαγή με τους Βρετανούς, υπάρχει κάποιο είδους μηδέα αναγνώριση γιατί με το hard Brexit ε, πώς θα εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία από την Βρετανική πλευρά. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Σημαντικό το ερώτημα αυτό. Η Σίλβια. Και εγώ ήθελα να ξέρω. Γιατί εδώ γίνεται λόγος για όσους είναι μέρη της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας, αλλά όχι της άλλης, γιατί ακόμα δεν ξεκίνησε Η άλλη ερώτηση αφορά αυτό που λέγαμε και πριν. Δηλαδή την εγγύηση αμοιβαιότητα αυτή τη αναγνώριση. Καταλαβαίνω πω είναι πολύ περίπλοκο το να σα ρωτήσω εάν ε, ισχύει, εφόσον υπάρξει Brexit. Όλα αυτά γίνονται εάν είναι εγγυημένη η αμοιβαιότητα. Αν υπάρχει αναγνώριση των ε, βαθμών και των πόρων. Οι πόροι φαίνεται πως καλύπτονται από τον προπολογισμό του 19 που το καλύπτει το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πόροι για το 19, εάν υπάρξει hard Brexit κάτι τέτοιο δεν θα γίνει. Δηλαδή αναγνωρίζουμε μόνο το χρόνο για εκείνους που έχουν ήδη ξεκινήσει. Αυτό σημαίνει πως καλύπτεται ήδη από τους πόρους ε, που καλύπτει το Ηνωμένο Βασίλειο ή πρέπει και εκεί να ε, εγγυηθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δρογεύσκη. Uczestniczyłem w imieniu pani przewodniczącej w ostatnim spotkaniu. Σας ευχαριστώ. Εγώ συμμετείχα στην τελευταία σύσκεψη με τον Μισελ Μπαρνιέ στο όνομα της Προέδρου και τότε ρώτησα κάτι για το Εράσμος ΣΥΝ. Θα πρέπει να πούμε καταρχάς ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να διατηρήσει το έρασμο Plus. Για μας αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από πλευρά τη Βρετανία, λοιπόν δεν υπάρχει θέληση να βγουν από αυτό το πρόγραμμα αλλά για να διευκρινιστούν τα θέματα τα νομικά. Εάν υπάρξει συμφωνία αυτό θα προχωρήσει. Αν όχι και έχουμε μια μεταβατική περίοδο με κάποιες δεσμεύσεις, ο Μισελ Μπαρνιέ είπε ότι κατά τη μεταβατική περίοδο δεν θα υπάρξει πρόβλημα για το πρόγραμμα Erasmus ε, Plus, γιατί θα είναι στη τελική του φάση. Εάν όμως ε, ε, γίνει hard Brexit, δηλαδή χωρίς συμφωνία, χωρίς μεταβατική περίοδο για τα διάφορα νομικά ζητήματα, τότε ποσοστώσεις, τελωνία κτλ λήψη σε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι στοιχείο μιας πρότασης για τη διατήρησή του στη πιο δύσκολη φάση του Brexit. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά τα όσα είπε η κυρία Διευθύντρια, εμείς προτείνουμε μια λύση χωρίς να κλείσουμε την πρόταση αυτή σε χρονικό πλαίσιο για να δούμε δηλαδή αν θα υπάρξει συμφωνία. Ωστόσο υπάρχει σοβαρό ζήτημα στο οικονομικό θέμα, γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θέλει να αποφύγει την οικονομική συμβολή του. Μπορείτε αυτό να μας το επιβεβαιώσετε. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνω. Αυτό, αυτή η πρόταση που έχουμε εδώ είναι ε, μια πρόταση μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία, που γίνει δηλαδή σκληρό Brexit. Brexit χωρίς συμφωνία δηλαδή. Όλα τα άλλα ενδεχόμενα είναι άλλη υπόθεση. Είτε δηλαδή ε, έχουμε μια συμφωνία για το τι θα γίνει μετά το 2020, ή μέχρι το 2020, μετά το 2021 κτλ. Δηλαδή μιλάμε για την περίπτωση που στις 29 Μαρτίου υπάρχει σκληρό Brexit και έχουμε ή 7.000 ε, άτομα ή 14.000 άτομα εδώ ή εκεί που έχουν μείνει ξεκρέμαστα. Δηλαδή τι κάνουμε με αυτούς στην περίπτωση αυτή. Αυτό δηλαδή αφορά η 7000 ατομα η 14000 ατομα εδω η εκει που εχουν μεινει ξεκρεμαστα δηλαδη τι κανουμε με αυτου στην περιπτωση αυτη αυτο δηλαδη αφορα η προταση που μας έχει υποβάλει. κυρία Μπίλντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέμε και ξαναλέμε ότι το Erasmus Plus είναι η μεγάλη επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε τόσο ικανοποιημένοι που σχεδόν όλα τα μέλη της Επιτροπής μας είναι υπέρ της διπλασιασμού του προπολογισμού αυτού του προγράμματος. Το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετείχε σε αυτή την επιτυχία γιατί είναι από τις πιο ε, επιθυμητούς προορισμούς. Ε, το 2015 και 2016, 126.000 φοιτητέ φοιτητές από ολόκληρη την Ευρώπη ε, ε, σπούδασαν εκεί, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο μόνο 14.000 φοιτητέ έστειλε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θα πρέπει να σημειώσουμε ποιε θυσίε κάνουν οι Βρετανοί, γιατί, γιατί οι φοιτητέ οι Ευρωπαίοι ε, πληρώνουν τα ίδια ποσά με τους Βρετανούς φοιτητές, ενώ οι τριτοκοσμικοί, τριτο, μάλλον, οι φοιτητές τρίτων χωρών πληρώνουν τα διπλάσια και τα τριπλάσια. Εφόσον ε, δεν είναι μέρος του έρασμους ε, το, ε, τα Βρετανικά Πανεπιστήμια, τότε το Κοινοβούλιο θα πρέπει να, να, να αποκομίσει τα συμπεράσματα των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος, αλλά και να εκδικηθεί για μια τέτοια σύγκρουση. Θα είναι όμως αυτό αντιφατικό με το μήνυμα της φιλίας των λαών που είναι στην πηγή ε, και στη ρίζα της Ένωσης. Το Ηνωμένο Βασίλειο έρχεται δεύτερο μόλις πίσω από τη ΣΥΠΑ. Ακόμα και αν τα δίδακτρα είναι εξαιρετικά ψηλά σας, καλό να σκεφτείτε τις συνέπειες. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο αποκλειστεί από το έρασμος Plus, όπως τρέφει τα νότα στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης. Αν λοιπόν αποκλειστεί το Ηνωμένο Βασίλειο, για, τότε γιατί θα συνέχιζε η Τουρκία ας πούμε, να είναι μέρος του έρασμος, ενώ δεν, έχει, δεν είναι καν υποψήφια ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δείχνει οι δηλώσεις και η συμπεριφορά του Ερντογάν. Κυρία Σόιντροπα, ευχαριστώ. Εγώ ε, αρχικά θέλω να αντιδράσω στην Γαλλίδα συνάδελφο. Με συγχωρείτε, αλλά αυτή η συζήτηση δεν έχει να κάνει με κανέναν αποκλεισμό της Μεγάλης Βρετανίας, διότι δεν έχουμε αποφασίσει εμείς για το Brexit. Εμείς πρέπει να αντιδράσουμε στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι φοιτητές οι φοιτητέ μας, οι Ευρωπαίοι φοιτητέ που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Ε, ευχαριστώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίως ε, έχω την ίδια ερώτηση όπως είχε και η Σαμπίνα. Πώς θα διαπραγματευτούμε για την κατάσταση για τους φοιτητές μας που θα παραμείνουν στην ε, Βρετανία στη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί 7.000 φοιτητές που βρίσκονται εδώ, από ό,τι κατάλαβα, θα τους ε, υποδεχτούμε Τι θα κάνει όμως η Μεγάλη Βρετανία για τους φοιτητές τους υπόλοιπους Ευρωπαίους που θα παραμείνουν στην Μεγάλη Βρετανία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ. Κυρία Άριξον. έχετε τον λόγο για να δώσετε απαντήσεις σε αυτά τα φλέγοντα ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σα. Καταρχάς, προς διευκρίνηση. Το αναφέρατε κι εσείς και η Πρόεδρος. Φυσικά, αν είχαμε συμφωνία, δεν θα χρειαζόμασταν ε, αυτόν, αυτήν εδώ την πρόταση. Θα τελείωναν τα προγράμματα όταν τελείωνε και το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Στην περίπτωση όμω, που αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς συμφωνία, οι δραστηριότητε οι οποίε χρηματοδοτούνται από το Erasmus Plus δεν θα είναι πλέον επιλέξιμε για χρηματοδότηση. Είναι λοιπόν μία λύση έκτακτη ανάγκη για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και με τον κανονισμό θέλουμε αυτές οι δραστηριότητες ε, για τις οποίες έχει ήδη ε, υπάρξει συμφωνία θα συνεχίσουν να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση. Δηλαδή δεν θα χρειαστεί να διακόψουν οι συμμετέχοντες τις σπουδές τους ή την άσκησή τους και να γυρίσουν πίσω. Θέλει λοιπόν η συμφωνία να διασφαλίσει την ολοκλήρωση του προγράμματος για τους συμμετέχοντες. Αμφίδρομα. Τώρα, όσοι Ευρωπαίοι πολίτε βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και όσοι Βρετανοί πολίτε βρίσκονται εδώ το κάνουν αυτό κατόπιν συμφωνιών που έχουν υπογραφεί. Δεν χρειάζεται λοιπόν καινούριε διαπραγματεύσεις. Εφόσον ε, τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός θα διασφαλίσει την ομαλή συνέχεια των προγραμμάτων μέχρι να ολοκληρωθούν. Δεν υπάρχει λοιπόν ανάγκη να γίνουν νέες διαπραγματεύσεις. Στην ουσία παρατείνουμε την περίοδο πληξιμότητας. Ε, συγγνώμη που σας διακόπτω, λέει πρόεδρος. Αλλά τι γίνεται αν ας πούμε οι Βρετανοί πούν, για παράδειγμα, πως ε, οι συμμετέχοντες σε προγράμματα στο έδαφος μας ε, χρειάζονται άδεια παραμονής. Και τι γίνεται όταν, ας πούμε, ένα συμμετέχον είναι πολίτης τρίτης χώρας, δηλαδή όχι ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, εντάξει, ας πούμε, ένας Τσέχος, ένας ε, Γερμανός, ένας Ιταλός που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, ίσως χρειαστεί βίζα για να μείνει στη χώρα. Ε, ασφάλιση. Ναι, η κυρία Φερχάιν διακόπτη. Πώ θα ρυθμιστούν λοιπόν αυτέ οι λεπτομέρειε. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του. Δεν μπορούμε εμεί να αποφασίσουμε κάτι για, τους, ε, για την προστασία των ε, Ευρωπαίων φοιτητών στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρί να συμφωνήσουν οι Βρετανοί. Δεν γίνεται το ένα άλλο. Τι γίνεται με τις μονάδες θα αναγνωριστούν από τα ευρωπαϊκά ιδρύματα. πώς θα προστατευτούν οι Βρετανοί φοιτητέ εδώ. Όμως η ερώτησή μου αρχικά είχε να κάνει με του, την προστασία των Ευρωπαίων φοιτητών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν, τι θα γίνει ας πούμε αν δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδέ τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια όμως ε, δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Γιατί είπατε κι εσείς ότι υπάρχουν ορισμένες δεσμεύσεις από τους Βρετανούς να μην διώξουν σπουδαστές οι οποίοι βρίσκονται εκεί στο πλαίσιο της κινητικότητας. Βέβαια αυτό δεν είναι δική μου αρμοδιότητα και ίσως είναι κάτι με το οποίο θα μπορούσε να ασχοληθεί κάποιος άλλος, κάποια άλλη επιτροπή. Εμείς βέβαια προσπαθήσαμε να κάνουμε πολλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά υπάρχει και διακυβερνητική συνεργασία με βάση της, ε, την ε, Μπολόνια. Υπάρχει δηλαδή το σύστημα μονάδων, διδακτικών μονάδων. Υπάρχει η συμφωνία για την αναγνώριση που είναι διακυβερνητική. Δεν νομίζω να υπάρχει λοιπόν θέμα μη αναγνώρισης προσόντων, περίοδων σπουδών στο εξωτερικό ή μονάδων, ας πούμε. Τώρα, για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είχατε μια ερώτηση και θα πω ότι η προσέγγιση σίγουρα είναι άμεση και πολύ περιοριστική. Αυτό σημαίνει το νέο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και λέω νέο ναι, γιατί πρόσφατα εγκρίθηκε ο κανονισμός, είναι κάτι νέο και το σημαντικό είναι να δούμε ότι βρίσκεται ακόμα σε πρώτο στάδιο. Οι περισσότεροι εθελοντές δηλαδή υπάρχονται στο Erasmus Plus και καλύπτονται από αυτήν την πρόταση. Ωραία. Προφανώς πολλά από τα ερωτήματα που προκύπτουν δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε. Απλώς θα ήθελα παρακαλώ να τα μεταβιβάσετε στην Κομισιόν ότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς τους νέους που είτε βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 30 Μαρτίου είτε είναι Βρετανοί και βρίσκονται κάπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 30 Μαρτίου για αυτούς να τους δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ασφαλές, νομικά ασφαλές. Όχι μόνο για τις ε, υποτροφίες τους ή για τα χρήματα που, θα τους, ε, που πρέπει να πάρουν από το Εράσμους, αλλά ε, ας πούμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δικαιώμα, δικαιώμα ε, παραμονής, για να μπορούν να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους απελάσουν από, την Ευρωπαϊκή, από, την, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ξέρω ότι σε αυτόν τον κανονισμό αυτό δεν μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Αλλά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εξασφαλίσουμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προσπαθήσει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσει ότι για αυτούς τους πολίτες, για αυτούς τους 21.000 νέους θα υπάρξει ασφάλεια δικαίου. Για να μην φοβούνται, να μην έχουν άγχος ότι αύριο θα καταλήξουν έξω από την πόρτα του σπιτιού τους, ότι θα τους διώξουν ή ότι δεν θα έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή οτιδήποτε. Ένα ερώτημα κρίσιμο. Σε... Υπάρχει αυτή η περίπτωση να μην υπάρξει συμφωνία. Παρόλο που είναι, δεν είναι πολύ δημοφιλής ε, περίπτωση, πάντα υπάρχει μια τέτοια περίπτωση το είχε καταλάβει από νωρί η Κομισιόν για το τι θα γίνει, ποια θα είναι η συνέπεια του κάθε σεναρίου. Υπάρχει, το, υπάρχει περίπτωση να μην γίνει Brexit, υπάρχει περίπτωση Brexit με συμφωνία, υπάρχει και η περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία. Η Κομισιόν τώρα ασχολήθηκε με τα ερωτήματα αυτά ή το έχετε από καιρό στο νου σας. Η κυρία Σόντροβα. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Ξέρω ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε εδώ, εφόσον δεν ξέρουμε ότι θα διασφαλίσουμε τα ίδια δικαιώματα για τους Βρετανούς με αυτά που θα έχουν οι Ευρωπαίοι φοιτητέ. Πρέπει να υπάρχουν ίδια δικαιώματα και για τους Βρετανούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι και οι δικοί μας οι οι Ευρωπαίοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα έχουν το ίδιο καθεστώς. Θα μπορούν να απολαμβάνουν των ίδιων δικαιωμάτων. Πρέπει να υπάρχει μια αμοιβαία συμφωνία λοιπόν ως προς αυτό με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και νομίζω ότι οι Βρετανοί θα το κατανοήσουν αυτό. Αν τους το ξεκαθαρίσετε και τους το εξηγήσετε ρητά, θα πρέπει να έχουμε ως βάση μια κοινή συμφωνία για να γίνουν όλα αυτά που θέλετε. Ευχαριστώ. Πολύ σημαντικά τα ερωτήματα που έχετε θέσει, αλλά το πεδίο εφαρμογή αυτού του κανονισμού δεν μπορεί να τα ρυθμίσει όλα αυτά τα θέματα. Οπότε, ίσως να πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε σε κάποιο διαφορετικό πλαίσιο. Αυτό που προσπαθεί να κάνει ο κανονισμός, πέραν των άλλων μέτρων που μπορεί να χρειαστούν, είναι να εξασφαλίσει ότι τα, οι τρέχουσε δραστηριότητε κινητικότητα θα μπορέσουν να, να συνεχίσουν να είναι επιλέξιμε για χρηματοδότηση, γιατί όλες αν δεν έχουμε αυτόν τον κανονισμό και όλε οι υπόλοιπε προποθέσει τηρούνται, δεν θα μπορούν να συνεχίσουν οι άνθρωποι που είναι στο, Erasmus, στο πρόγραμμα Erasmus τι δραστηριότητέ του. Εντάξει, λοιπόν, καταλάβαμε. Τα προγράμματα αυτά, μάλλον, τα προβλήματα συγγνώμη, αυτά, μάλλον επί τόπου θα πρέπει να λυθούν. Αυτό που μπορούμε εμεί να ρυθμίσουμε σε αυτόν τον κανονισμό θα ρυθμιστεί και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Ε, ευχαριστούμε και πάλι την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ να διαβιβάσετε ωστόσο τις ανησυχίες που έχουμε για όλα τα υπόλοιπα θέματα για να μπορέσει ίσως η Κομισιόν να μας ξεκαθαρίσει τι γίνεται είτε και γραπτός να μας δώσει κάποιες απαντήσεις για να, να μπορείτε να μας διασφαλίσετε ότι θα υπάρξει σαφήνεια για να εξασφαλίσουμε νομική ασφάλεια για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ωραία. Λοιπόν, το κλείνουμε το σημείο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αριξόν που ήσασταν εδώ σήμερα και μας ξεκαθαρίσετε λίγο το τοπίο και περνούμε κατευθείαν στην συνεδρίαση των συντονιστών. Να δούμε τι θα γίνει σε τεχνικό επίπεδο γιατί μόλις δύο εβδομάδες έχουμε για να μπορέσουμε να τα προωθήσουμε τα θέματα αυτά από εκείνο με το Συμβούλιο και σίγουρα αυτό είναι μια μικρή πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν στους συντονιστές όλα αυτά και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε και καλά συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ σήμερα και θα τα πούμε την επόμενη φορά. So, dann wären wir am Ende der Tagesordnung an. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της ημερήσιας διάταξης. Δεν υπάρχει τίποτα στα διάφορα. Μόνο να σας ενημερώσω ότι η επόμενη συνεδρία θα λάβει χώρα στις 20 Φεβρουαρίου, Τετάρτη, από τις 9 ως τις 12.30 και από τις 3 ως 6.30 και 21 Φεβρουαρίου